Ο Πρόεδρος. Αρχίζουμε αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε. We will start in 30 seconds. Αρχίζουμε σε μισό λεπτό. 30 δευτερόλεπτα για την ακρίβεια. Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορούμε να αρχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Είναι μια διάσκεψη πάρα πολύ σημαντική, κοινή διακοινοβουλευτική συνάντηση. Είναι πάρα πολύ μεγάλη σημασία για όλους, για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένωση και Δυτικά Βαλκάνια. Έχουμε σε 21 γλώσσες ταυτόχρονη διερμηνία. Όπω γίνεται σύντομα στι συνεδριάσει μα και θα ζητήσω συγγνώμη από του Μαλτέζου συναδέλφου, διότι Μαλτέζικα α, δεν προβλέπονται. Συνήθω έχουμε 22-23 γλώσσε προ τι οποίε γίνεται η διερμηνία, και αυτό γίνεται στις ε, κοινοβουλευτικές επιτροπές και στις ε, ολομέλειες, στις ε, όμως αλλά έχουμε όμως και κάποιους που δεν έχουμε συνήθως κροατικά, βοσνιακά, σερβικά και μαυροβουνιακά, μακεδονικά, λέει ο πρόεδρος, και αλβανικά. Εσείς επομένως, κατά βούληση, θα επιλέξετε τον διάβλο διερμηνίας, τον οποίο επιθυμείτε για να ακούτε την γλώσσα της αρεσκίας σας. Πρέπει να αρχίσω με το να εκφράσω τη χαρά μου γιατί κάναμε αυτή τη διοργάνωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και νομίζω ότι έτσι τονίζεται η δέσμευσή μας από πλευρά Ευρώπη προ τα Δυτικά Βαλκάνια, που είναι μια υπόθεση πάρα πολύ σημαντική για όλου και πρώτα-πρώτα να, να ευχαριστήσουμε τον ε, πρόεδρο Κόβερ, ο οποίος θα συμπροεδρεύσει και είναι ο πρόεδρος της ε, Εθνοσυνέλευσης της Ουγγαρίας. Ευχαριστώ επίσης τους αδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια που έχουν προσέλθει και επίσης τους προέδρους των ε, κοινοβουλίων της περιφέρειας με την οποία σήμερα συναντώμε δηλαδή τα Δυτικά Βαλκάνια. Όλοι αυτοί που ήρθαν σήμερα εδώ, ούτως ώστε να συνεργαστούμε και έτσι να στρώσουμε το δρόμο α, αυτή την πορεία μας προς μια ενωμένη Ευρώπη. Και επίσης βέβαια τελευταία και σημαντική είναι οι συνάδελφοί μου εδώ από το Ευρωκοινοβούλιο ε, εσάς δεν σας καλωσορίζω γιατί είσαστε κι εσείς ε, συν οικοδεσπότες μαζί μου. Πάντω χαίρομαι πάρα πολύ που όλοι βρεθήκαμε εδώ και έχουμε μπαίνει σε αυτέ τι κοινέ ε, διακοινοβουλευτικέ συνεδριάσεις που αποτελούν το πλαίσιο τη διακοινοβουλευτική συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια ε, συνεργασία αντιπροσωπευτική, κλασική, πάρα πολύ σημαντική και αποκτά όλο ένα και περισσότερη σημασία τώρα με την συνθήκη τη Λισαβόνα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, έχει δεσμευτεί προ τα Δυτικά Βαλκάνια, προ του λαού από τότε που είχαμε την διάσκεψη κορυφή του 2003 στην Θεσσαλονίκη. Τόσο παλιά. Πάρα πολύ σημαντική εκείνη η συνάντηση για την περιοχή εκείνη, διότι ε, καταργήσαμε τις θεωρίες διαβατηρίων για, για Μαυροβούνιο, ε, Σερβία και για την πρώην κοινωνική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Επίσης, ε, εγκρίναμε να γίνουν αντίστοιχα διαδήματα για Βοσνία-Ριζεγοβίνη, και μόλις μπορούμε να έχουμε όλες τις σχετικές προϋποθέσεις τότε θα πρέπει να καλύψουμε και το κρυσφοπέδιο οπότε και αυτοί χωρίς το διαβατήριο να μπορούν να ταξιδεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης Σερβία, Κροατία είναι οι χώρες οι οποίες έχουν κάνει κάποια πολύ σημαντικά βήματα προς την ολοκλήρωση οι πρόεδροι Τάντιτς και Γεσίποβιτς διότι έτσι δείχνουν το πόσο, πόσο ε, έχουν λάβει τέτοιου είδους ε, πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, κοινή πορεία, ενώ πριν ήταν ε, εχθροί, τώρα θα μπορέσουν να συνεπάρξουν ειρηνικά και θα είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση για την ευημερία, την ειρήνη στην περιοχή, κάτι το οποίο επίσης είναι κλασικό όσον αφορά την Ευρώπη. Θα πρέπει επίσης να μην ξεχνούμε τι έγινε τι τελευταίε δεκαετίες. Ε, άλλωστε μην ξεχνούμε τη συμφιλίωση, την γάλλο-γερμανική, ε, την Πόλωνο-Γερμανική και άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Πολύ σημαντικά φαινόμενα όλα αυτά. Επίσης, φέτος μόλις το Μαυροβούνιο εχρήστη υποψήφια χώρα. Και αυτό γιατί καταβάλλονται όλες οι προσπάθειες τόσο ώστε να, να μπει στην τελική ευθεία για την προσχώρηση. Οπότε όλα αυτά είναι καλά μαντάτα για όλη την περιφέρεια για όλη την Ευρώπη και όχι μόνο για αυτές τις δύο χώρες παραλαμβάνω διότι έχουμε πάρα πολλά τέτοια μηνύματα ενθαρρυντικά υπάρχουν ένα σωρό ε, προκλήσεις και θα πρέπει επομένω όλα αυτά να τα συζητήσουμε, να ανακαλύψουμε τα θέματα που υπάρχουν και όλε οι χώρε έχουν παρόμοια προβλήματα στην περιοχή εκείνη. Θα πρέπει δηλαδή να προβούν σε κάποιε μεταρρυθμίσει ε, στη δικαιοσύνη, να κατομιλήσουν την ε, διαφθορά. Θα πρέπει να συνεχιστεί η συνεργασία, η συμφιλίωση. Ε, και άλλωστε πρόσφατα μας προβλημάτισε ιδιαίτερος το ότι υπήρξαν ε, κάποια δείγματα πολιτικής ασταθείας στην περιοχή. Επίσης θα πρέπει να σας υπενθυμίσουμε ότι η Βοσνία Ερζεγοβίνη από τότε που έγιναν οι εκλογές τον Οκτώβριο δεν κατάφερε να σχηματίσει η κυβέρνηση και επίσης ε, όσον αφορά την, την, την Αλβανία και εκεί έχουμε κρίση οπότε θα πρέπει να δούμε το ότι κάθε φορά που δεν σχηματίζεται η κυβέρνηση μετά από εκλογέ σταματούν οι μεταρρυθμίσει. Και έτσι προχωρούν και οι διαπραγματεύσει. Πάντω, οπωσδήποτε ακολουθούνται οι δημοκρατικέ συνταγέ και μέθοδοι, ούτω ώστε να επιληθούν τα προβλήματα. Τίποτα καλύτερο δεν υπάρχει από τη δημοκρατία για τέτοιου είδου ε, λειτουργία που είναι η συνήθι λειτουργία εδώ των θεσμικών οργάνων. Έτσι κάνουμε και έτσι νομοθετούμε. Επομένω, είναι πάρα πολύ σημαντικό όλοι οι πολιτικά εμπλεκόμενοι, οι πολιτικοί παίκτε να ξεπεράσουν όσα του διχάσουν και να υπάρξει επικοδομητική συνεργασία μεταξύ κυβέρνηση αλλά και αντιπολίτευση. Να, μια πάρα πολύ σημαντική πρόκληση πέρα από την ε, περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων διότι έχουμε την λεγόμενη κόποση τη διεύρυνση. κάτι το οποίο σοβεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση Επομένω, θα πρέπει να πείσουμε του Ευρωπαίου όσον αφορά τα υπέρ τη διεύρυνση. και όταν λέμε τους πολίτες εννοούμε του πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και πρόκειται για μια πτυχή πάρα πολύ σημαντική <coughs> για την μέλουσα πορεία της διεύρυνσης γιατί μέλουσα διεύρυνση για όλα τα βαλκανικά κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως, Έχουμε δύο ομάδες που θα αρχίσουν να συνδυάζουν τότε τις 5 η ώρα και θα ζητήσουν σημαντικά ζητήματα. Η πρώτη ομάδα θα ζητήσει τα της συνεργασίας όσον αφορά την ελευθερία, την δικαιοσύνη και την ασφάλεια. Αυτά έχουν ε, αποτυπωθεί στη συνθήκη της Λισαβόνας και επίσης έχουμε μια δεύτερη ομάδα εργασίας που θα ασχοληθεί με την ε, ένταξη, την κάλυψη των πολιτών σε σχέση με την πολιτιστική πολυμορφία. Είναι κάτι το οποίο αφορά την Ευρώπη όλη και όχι μόνο τα Βαλκάνια, διότι θα πρέπει πάντοτε να θυμόμεθα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά θέματα αυτά όσον αφορά την ε, ένταξη των πολιτών και την ε, κάλυψή τους από αυτήν την πολιτιστική πολυμορφία. Ε, επομένως έτσι μοιραζόμαστε κάποιες ιδέες και όσο πιο νυχτές είναι οι συζητήσεις μας, τόσο πιο εύκολα θα καταφέρουμε να επηρεάσουμε την σύνοδο, την σημαντική του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Ιούνιο. Η εμπειρία μας λέει ότι θα είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά πάντως πρέπει να σας πω ότι επίσης αυτή η δύσκολη πορεία που έχουμε διανύσει άξιζε να γίνει και κατά αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να αναδείξουμε τις ευρωπαϊκές προοπτικές των Δυτικών Βαλκανίων, την ευρωπαϊκή πραγματικότητα, ε, την, την συνύπαρξη ε, μαζί τους στο ή δυνατόν εγγύς μέλλον. Συνάδελφοι, θα πρέπει να σας πω ότι ξεκινούμε τώρα την ημερησία διάταξη την οποία έχετε λάβει. Ξέρετε τι θα έχουμε κάνουμε σήμερα ε, και αύριο. Αύριο θα έχουμε εδώ τον Πρωθυπουργό Όρμπαν της ε, Ουγγαρίας που ασκεί την Προεδρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το εξάμεινο και επίση θα έχουμε και τον Ζωσέ Μανουέλ Μπαρόσο, τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οπότε θα έχουμε αυτούς τους υψηλούς προσκεκλημένους μας αύριο το πρωί. Σήμερα όμως, σήμερα όμως με μεγάλη μου χαρά θα δώσω την σκητάλη, θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο που προεδρεύει. Mr ο επομένω επομένως της ε, Ουγγρικής Εθνοσυνέλευσης ε, Λάσλο Κέβερ. Λάσλο, έχεις το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σας απευθύνω ένα φιλικό χαιρετισμό σε αυτήν την ε, μεικτή κοινοβουλευτική συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ουγγρικής Εθνοσυνέλευσης. Κύριε Μπούζεκ, σας ευχαριστώ όλος ιδιαίτερως ε, για την αγαστή συνεργασία που είχαμε μέχρι στιγμής. Όλες αυτές οι μικτές συνεδριάσεις εντάσσονται σε ένα γενικότερο πλαίσιο, δημοκρατικό πλαίσιο, που μας επιτρέπει να εξετάζουμε τα πιο επίκαιρα, δύσκολα θέματα που μας απασχολούν. Δεν έρχομαι εδώ εκπροσωπώντας την Ουγγρική Προεδρία. Ερχόμαστε εδώ πέρα για να συζητήσουμε ένα θέμα που είναι σημαντικό για ολόκληρη την Ευρώπη. Η Ευρώπη επιθυμεί να διατηρήσει την ταυτότητά της, τον πολιτισμό της, την ειρηνική συμβίωση των λαών της αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι πάρα πολύ σημαντικό να κινούμεθα μέσα σε ένα ειρηνικό, φιλιρινικό πνεύμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε τα νέα κράτη-μέλη που προσχώρησαν, ε, κάποια το 2004, κάποια άλλα το 2007 Ελπίζουμε να μην έχει σημάνει το τέλος της διαδικασίας διεύρυνσης και ελπίζουμε ότι οι διάφορες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων σύντομα θα εισέλθουν στην Ένωση. Η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης έχει ιδιαίτερη σημασία Ο στόχος είναι η ολοκλήρωση ολόκληρης της ε, γυραιάς Υπήρου, σημαίνοντας ε, το πραγματικό τέλος ε, της βίας και του ψυχρού πολέμου που γνωρίσαμε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. θα εξετάσουμε δύο διαστάσεις του ζητήματος, ε, η ελευθερία, η ασφάλεια, η δικαιοσύνη, ο έλεγχος των συνόρων, η μεταναστευτική πολιτική, πολιτική θεωρήσεων, πολιτική συνεργασία, αστυνομική συνεργασία, δικαστική συνεργασία. Και η πορεία των χωρών των Δυτικών ε, Βαλκανίων θα καταδείξει μία ακόμη φορά τη σημασία της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Προσπαθήσαμε από πλευράς μας να ενισχύσουμε τη διαδικασία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες με διάφορες εθνοσυνελεύσεις από χωρών Δυτικών Βαλκανίων θα ανταλλάξουμε τις εμπειρίες μας και θα συνεργαστούμε προφανώς και σε διοικητικό επίπεδο. Αυτό θα απαιτήσει συντονισμό των δράσεων των Προέδρων των Κοινοβουλίων αυτών των χωρών. Ε, η περιοχή αυτή της Ευρώπης ε, διέρχεται μια περίοδο δημοκρατικής μεταρρύθμισης Έχουμε ήδη ε, ανταλλάξει απόψεις για αυτό το θέμα το Φεβρουάριο, παραδείγματος χάρη, με τους προέδρους των Εθνοσυλλελεύσεων, στην κοινή μας διάσκεψη ε, και δεν είναι η μόνη το 2003, το 2005, το 2007 ε, οργανώθηκαν τέτοιες διασκέψεις, η τελευταία ήταν στη Βουδαπέστη και το φθινόπωρο θα οργανώσουμε και άλλη μία διάσκεψη όπου θα καλέσουμε τους Προέδρους των Εθνοσυνελεύσεων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Θα ήθελα να προσθέσω ότι θα συμπροεδρεύσουμε με τον Πρόεδρο Μπούζεκ, με μεγάλη τιμή για μένα. Ο κύριος Μπαμπίτσκ θα μας κάνει μια παρουσίαση για την οικονομική ολοκλήρωση. Πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό το να καταλάβουμε πως ε, δεν έγκυται μόνο στην προσχώρηση στην Ένωση η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Σχετίζεται επίσης με την περιφερειακή συνεργασία και γι' αυτό το λόγο είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διατηρούμε οικονομικές και πολιτιστικές σχέσεις σε αυτή την περιοχή της Ευρώπης. Ο στόχος δεν είναι να καταστούν πιο εύρωστες οι οικονομίες μας, ε, ε, μπορούμε με διάφορους τρόπους να υποφεληθούμε από την πρόοδο που έχει ήδη σημειώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ και προσβλέπω στον επικοδημητικότατο διάλογο που θα έχουμε. Πρόεδρος Μπούζεκ, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα... Να σας πω ποιοι θα είναι οι κανόνες για τη συζήτηση. Ο συνάδελφος Κέβελ μας τα είπε προηγουμένω. Έχουμε δύο φιλοξενούμενους ομιλητές, καλωσορίζουμε. Τον κύριο Λούκα Μπέμπιτς από το Κρατικό Κοινοβούλιο. Πριν μερικέ μερικές ώρες συναντηθήκαμε. Συζητήσαμε πολλά. Και η κυρία Σόνια Μπιζέρκο, επικεφαλής της Επιτροπής του ΕΣΥΝΚΙ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Σερβία. Να σε εξηγήσω το επόμενο σημείο. Προσυζήτηση. Θα γίνει ζωντανή συζήτηση Θέλουμε να παρέμβετε σε αυτή τη συζήτηση και να το ζητήσετε μέσω του, του εντύπου που λέει ζητώ χρόνο αγόρευσης, αγόρευσης την Τετάρτη στην Ολομέλεια της μικτής αυτής κοινοβουλευτικής συνέλευσης. Σας δώσαμε τέτοιο έγγραφο. Τέτοια έντυπα έχετε. Μπροστά σας έχετε τέτοιο έντυπο. Συμπληρώστε το λοιπόν αν θέλετε το λόγο και βάσει των αιτήσεων αυτών που θα λάβουμε θα συντάξουμε έναν κατάλογο ομιλητών. Θα το ετοιμάσει δηλαδή η γραμματεία της διάσκεψης. Ξεκινήστε λοιπόν τώρα. Ετοιμάστε ένα αίτημα αν θέλετε να πάρετε το λόγο. Και δεύτερο σημαντικό θέμα. Ο χρόνος αγόρευσης είναι τρία λεπτά για τον καθένα από εσά που συμμετέχετε στη συζήτηση. Και τρίτον, λίγο περίπλοκο αυτό, αν θέλετε να παρέμβετε και να ρωτήσετε, να θέσετε ένα ερώτημα, οποιοδήποτε. Από οποιοδήποτε ομιλητή που μιλάει τρία λεπτά, σηκώνεται γαλάζια κάρτα. Και αυτή θεωρείται παρέμβαση της γαλάζιας κάρτας. Μπορείτε να αποβάλλετε σύντομο ερώτημα ή να πείτε κάτι για 30 δευτερόλεπτα. Και μετά θα απαντηθεί από τον ομιλητή και αυτό θα έχει χρόνο 30 δευτερόλεπτα για να απαντήσει. Έτσι θα είναι και πιο ζωντανή και ζωηρή συζήτηση. Συνεννοούμαστε έτσι. Καταλάβατε τη διαδικασία αυτή που σας περιέγραψα με τη γαλάζια κάρτα. Αν θέλετε να θέσετε οδήποτε ερώτημα προς τον ομιλητή που μόλις τώρα έχει το λόγο, τη στιγμή που έχει το λόγο, σηκώνετε τη γαλάζια κάρτα. Ξεκινάμε λοιπόν από την πρώτη παρέμβαση η βασική παρέμβαση του κ. Λούκα Μπέμπιτς, που είναι ο πρόεδρος του Κρατικού Κοινοβουλίου. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητέ Πρόεδρε, κύριε Μπούσεκ, του, κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Ουγγρικής Εθνοσυνέλευσης, κύριε Κβέρ, αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, με μεγάλη χαρά δέχτηκα αυτή την πρόσκληση να συμμετάσχω σε αυτή την μεικτή κοινοβουλευτική σύνοδο όπου έχω τη δυνατότητα παρουσία των υψηλότερων αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ενώσης να, περι... να πω μερικά πράγματα για την οικονομική συνεργασία στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η Κροατία και το Κρατικό Κοινοβούλιο εκτιμούν πολύ την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κατά τη διάρκεια των ενταξιακών διαπραγματεύσεων για την ένταξη της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις 16 Φεβρουαρίου είδαμε πιο έντονα την υποστήριξη μέσω του ψηφίσματος για την πρόοδο που πέτυχε το 2010 η Κροατία. Η υποστήριξή σας σημαίνει πολλά για μας και εφόσον περνάμε τώρα τα τελευταία μέτρα του μακριού δρόμου που ξεκίνησε την περασμένη δεκαετία. Ε, έτσι επιβεβαιώνεται η πεποίθησή μας ότι δεν είμαστε μόνοι σε αυτό το δρόμο και θα είναι πιο εύκολο για μας να πετύχουμε το στόχο ένα στόχο που θέλαμε να πετύχουμε, να τελειώσουμε τις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τέλος Ιουνίου φέτος. Για να πετύχουμε αυτό το στόχο υπάρχουν 7 κεφάλαια που θα πρέπει να κλείσουν και είμαστε δεσμευμένοι, θέλουμε να κλείσουν. Η επιτυχία των διαπραγματεύσεων των ενταξιακών είναι και επιτυχία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ενώσης και επιβεβαιώνει την προοπτική ε, που υπάρχει για άλλες χώρες να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύντομα θα τελειώσουν οι διαπραγματεύσει λοιπόν τη Κροατία για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκεί θα φανεί ποιο είναι ο πραγματικό προσανατολισμό των χωρών της, ε, των Δυτικών Βαλκανίων. Οι διαπραγματεύσει τη Κροατία και η όλη εμπειρία και οι ευρωπαϊκέ ε, προοπτικέ είναι μεγάλη ενθάρρυνση για μα. Η περιοχή και η περιφερειακή συνεργασία είναι στο επίκεντρο τη προσοχή τη εξωτερική πολιτική τη Κροατία. Βεβαίω είναι σημαντικό να έχουμε καλές ε, γειτονικές σχέσεις και σχέσεις εταιρικής συνεργασίας με όλες τις περιοχής είναι κάτι που μας επιτρέπει να συμβάλλουμε μακροπρόθεσμα στη δημιουργία μια, ενός χώρου ειρήνης, σταθερότητας και ευμαρίας στην περιφέρεια αυτή. Έτσι περαιτέρω με την εμπειρία και την αποκτηθήσα γνώση κατά συνταξιακές διαπραγματεύσει, η Κροατία είναι έτοιμη να υποστηρίξει χώρες της περιοχής στο δικό τους δρόμο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλες οι περιφερειακές μας δραστηριότητε και σε διμερές επίπεδο ε, και σε πολυμερή προγράμματα όπως το ΣΕΦΤΑ, όλες οι προσπάθειες που καταβάλουμε η ΣΕΦΤΑ που είναι η διαδικασία της συνεργασίας στην Ανατολική ε, Ευρώπη και το Συμβούλιο της Ανατολικής Ευρώπης είναι σημαντικό τμήμα των προσπαθειών στην εξωτερική μας πολιτική. Στην προσπάθεια λοιπόν ενίσχυσης της περιφερειακής συνεργασίας η νοτιοανατολική Ευρώπη αρχεί να κατανοεί και να στερνίζεται τις αξίες που υποστηρίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πλήρης η συνεργασία ε, και επεκτείνεται στο δομέα της δικαιοσύνης, αστυνομίας, άμυνας, καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος και διαφθοράς. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία αναφέροντας τους σημαντικότερους οικονομικούς δείκτες και συγκεκριμένα στοιχεία επί των οικονομικών συναλλαγών της περιοχής οι οικονομικές προπτικές των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης είναι πολύ διαφορετικές από ό,τι είχαμε μπροστά μας πριν από 10 χρόνια. Σήμερα είναι μια αγορά περίπου 20 εκατομμυρίων καταναλωτών και η συνεργασία σε αυτή την αγορά ε, δημιουργήθηκε ε, επί τη βάση της ΣΕΦΤΑ. Όλες οι χώρες της περιοχής είναι χώρες που είναι σε μεταβατική περίοδο με σχετικά χαμηλό ΑΕΠ κατά κεφαλήν, αλλά έχουν τεράστιες δυνατότητες για οικονομική ανάπτυξη. Οι αναπτυσσόμενες οικονομίες της περιοχής είναι ταυτόχρονα και οι πιο δυναμικές στην Ευρώπη και είναι από συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη. Οι χώρες της περιοχής είναι χώρος νέων επενδύσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση κυρίως επενδύσεις σε υποδομές και ενέργεια. Και αυτός ο τομέας, ο οικονομικός, σίγουρα θα είναι πιο ελκυστικός στους επενδυτές Ευρωπαϊκής Ενώσεως και σε επενδυτές από άλλες χώρες σε κάθε βήμα που ακολουθούμε προς την ένταξη. Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της περιοχής είναι η επίτευξη οικονομικής πρόοδου και η βιώσιμη ανάπτυξη που αποτελεί εχέγγυο της ειρήνης και της σταθερότητας. Πιστεύω ότι είμαστε στο σωστό δρόμο για να εκπληρώσουμε τους στόχους μας. Τα στοιχεία όσον αφορά το εμπόριο μεταξύ των χωρών της περιοχής αυτής της Ευρώπης επιβεβαιώνουν την οικονομική συνεργασία μεταξύ ε, της κάθε χώρας με τις γειτονικές χώρες. Το, 200, το 2010 το εμπόριο μεταξύ Κροατίας και χωρών της περιοχής ήταν στο ύψος 2,5 δις ευρώ περίπου 10% όλο του εμπορίου της Κροατίας με χώρες ε, στον υπόλοιπο κόσμο. Το εμπόριο της Κροατίας με άλλες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης όσον αφορά τις εξαγωγές και τις εισαγωγές είναι στο πλεόνασμα. Άρα εξάγουμε περισσότερα. Εξάγουμε 1,66 δισεκατομμύρια ευρώ και εισάγουμε 812 εκατομμύρια ευρώ. Και άλλος τομέας στον οποίο μπορούμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία είναι οι καλύτερες μεταφορές στην περιοχή. Η δημοκρατία της Κροατίας, σύμφωνα με τις δυνατότητες που διαθέτει, θα εξακολουθεί να κατασκευάζει τον πανευρωπαϊκό διάδρομο 5C στο τμήμα που περνά βέβαια από, το, από τη χώρα, από την Κροατία. Ετοιμαζόμαστε να φτιάξουμε μια κοινή γέφυρα μεταξύ Κροατίας, Βοσνίας και Ζεγοβίνης ε, που θα γεφυρώνει το ποτάμι Σάβα στο διάδρομο 5C και καλωσορίζουμε τις προσπάθειες που καταβάλλονται στην γειτονική Βοσνία Ζεγοβίνη όσον αφορά την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου στον προαναφερθέντα διάδρομο. Θα ήθελα να πω επίσης ότι μαζί με τους ιδεοδρόμους της Σερβίας και της Σλοβενίας, η Δημοκρατία της Κροατίας ε, καταβάλει προσπάθειες για την άρση τελωνιακών και διοικητικών φραγμών ούτως ώστε ο σιδηροδρομικός διάδρομος 10 να γίνει όσο το πιο δυνα, ε, πιο ανταγωνιστικός δυνατότητα. Έχουμε και το Τζάναφ που δίνει πετρέλαιο από την παγκόσμια αγορά στη Σερβία, στα δηληστήρια της Σερβίας και στα δηληστήρια της Βοσνίας ε, Ζεγοβίνης. Και από τη στιγμή που θα έχουμε περισσότερες δυνατότητες αποθήκευσης, η Τζάναφ θα μπορέσει να προσφέρει χώρους αποθηκευτικούς παραγόγων πετρελαίου για τις χώρες της περιοχής οι δυνατότητες ε, ανάπτυξης στον ενεργειακό τομέα είναι κάτι που βλέπουμε στην σύνδεση αγωγών φυσικού αερίου στην περιοχή. Σημαντικό βήμα σχετικά με αυτό το θέμα είναι η δημιουργία της ενεργειακής κοινότητας της Νοτιοδυτικής Ευρώπης. Θα ήθελα να πω επίσης ότι η Κροατία βλέπει να υπάρχει τεράστια ε, οικονομική δυνατότητα σε συνοριακά προγράμματα που εφαρμόζονται εντός στρατηγικής για το Δούναβι η πρωτοβουλία για την Αδριατική και για το Ιούνιο και άλλε πρωτοβουλίε. Τώρα, όσον αφορά την περιφερειακή συνεργασία, το Συμβούλιο Περιφερειακής Συνεργασία υποστηρίζει η Κροατία αυτού του είδου τη συνεργασία που εστιάζεται επί συγκεκριμένων έργων και τονίζουμε ότι πρέπει να συμμετάσχει όλοι, όλες οι χώρες της περιοχής θα πρέπει να συμμετάσχουν και θα πρέπει να παραμείνει αυτή η συμμετοχή και στο μέλλον μαζί με τη ΣΕΦΤΑ και άλλες, άλλες υποδομές και έργα υποδομών ε, θα ήθελα να τονίσω ότι τεράστιε δυνατότητε που υπάρχουν για περιφερειακή συνεργασία στην περιοχή του Δούναβη. Έχει μεγάλη σημασία για την περιοχή. Γι' αυτό με μεγάλο ενθουσιασμό η Κροατία υποστήριξε και συμμετείχε στην εκτέλεση της στρατηγικής του Δούναβη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως σαν ένα σωστό πλήρες πλαίσιο για συνεργασία στην περιοχή. Πιστεύει η Κροατία ότι τέτοια πολυδιάστατη προσέγγιση στην περιφερειακή συνεργασία δημιουργεί στέρεα θεμέλια για την ευμάρεια και τη σταθερότητα της περιοχής, στο σύνολό της. Ε, ιδιαίτερα σημαντικά μέσα για περιφερειακή πολιτική και σαν απόδειξη του ενεργού ρόλου της Κροατίας στην περιοχή ε, θα πρέπει να αναφέρουμε και τη διάσκεψη που διεξήχθη πρόσφατα στο Ντουμπρόβνικ ε, η διάσκεψη Ρον Μπράουν που έλαβε χώρα τον, 4 Απριλίου μέχρι 6 Απριλίου μια διάσκεψη για το εμπόριο και επενδύσεις μεταξύ ΙΠΑ και Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η περιφερειακή συνεργασία θα παραμείνει μία από τις προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής της Κροατίας και ξέρω που μπορώ να επιβεβαιώσω εδώ ότι η Κροατία θα συνεχίσει να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην εντατικοποίηση της περιφερειακής ανάπτυξης ενισχύοντας τις σχέσεις μεταξύ των χωρών της περιοχής και η προσπάθεια θα εδράζεται επί συνεργασίας εταιρικών σχέσεων και ενισχύσεως του πολιτικού διαλόγου και ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον πρόεδρο Μπέμπιτς. Επόμενος ομιλητής, η κυρία Σόνια Μπισέλκο, επικεφαλής της Επιτροπής Ελσίνκη για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στη Σερβία. Ευχαριστώ ε, κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, αγαπητοί φίλοι. Σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε να μιλήσω σε αυτή την κοινή μεικτή κοινοβουλευτική συνεδρίαση. Μου αρέσει η πρωτοβουλία αυτή γιατί η διαρκή συμμετοχή και το διαρκές ενδιαφέρον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην περιοχή είναι πραγματική πραγματικά βασικές προϋποθέσεις για την πρόοδο. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει φτάσει σε ένα σημείο σε ό,τι αφορά την δεσμεύση τη στην περιοχή, όπου προαπαιτείται μια διαφορετική στρατηγική προσέγγιση για τις χώρες αυτές, οι οποίες επί σειρά ετών προσπαθούν να πατήχουν τα κριτήρια για να καταστούν υποψήφιες χώρες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να τονίσω ότι τα ζητήματα τα οποία θα συζητηθούν στις ομάδες εργασίας ε, σε ό,τι αφορά τη συνεργασία στον τομέα της δικαιοσύνης αλλά και σε ό,τι αφορά την ενσωμάτωση των πολιτών, είναι πολύ βασικά για την ενσωμάτωση των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, προκειμένου τα θέματα αυτά να ειδωθούν με τη σωστή προοπτική, θα πρέπει να έχουμε μια σωστή ιδέα για την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, γιατί δυστυχώ κάποια από τα κράτη τη περιοχή ακόμη δεν πληρούν κάποιε βασικέ προποθέσει για την δημοκρατικό ε, την δημοκρατική ε, διεξαγωγή ε, και την σωστή σχέση με τους γειτονές τους. Τι συμβαίνει λοιπόν στην παρούσα φάση. Η Βοσνία εξακολουθεί να μπλοκάρεται από την ιστορική πολιτική της κρίση. Η Μακεδονία ακόμα δεν μπορεί να ξεκινήσει διάλογο με την Ελλάδα. Το, το ζήτημα αυτό που επηρεάζει την Μακεδονία επηρεάζει την εξέλιξη της Μακεδονίας στην περιοχή. Το ίδιο και με το Κωσυφοπέδιο. Παρόμοια κατάσταση. Το δικαστήριο της Χάγης επιβεβαίωσε την ανεξαρτησία του Κωσυφοπεδίου αλλά δεν άλλαξε τη στάση της Σερβίας έναντι στο Κωσυφοπέδιο. Η σχετική έκθεση για την εμπορία οργάνων επίσης έχει ε, βλάψει πολύ την δημόσια εικόνα της χώρας. Κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι υπάρχουν ε, δύο παράλληλες ε, διαδικασίες οι οποίες διεξάγονται εδώ η ενίσχυση του κράτους και η μετάβαση σε ένα πολυκομματικό ε, πολιτικό σύστημα και στην οικονομία της αγοράς. Και οι δύο διαδικασίες προχωρούν υπερβολικά ίσως αργά. Σε ό,τι αφορά την πρώτη διαδικασία, να έχουμε υπόψη ότι κάποια κράτη, όπως είπα, είναι ακόμα ευάλωτα και απειλούνται από τις εθνικές εντάσεις. Σε ό,τι αφορά την δημοκρατική μετάβαση, τον αυταρχικό χαρακτήρα, ο αυταρχικός χαρακτήρας των ε, χωρών εξακολουθεί να επικρατεί παρά το πολυκολματικό σύστημα. Κάποια από τα παλιά επιτεύγματα επισκιάζονται από αρχαϊκές εθνικές, εθνικιστικές ιδεολογίες. Υπάρχει μια ισχυρή αντίσταση στην οικοδόμηση ενός συστήματος πλουραλισμού οικονομικού και μιας ε, ελεύθερης αγορής. Κυρίες και κύριοι, ένα από τα βασικά προβλήματα είναι η στάση της Σερβίας έναντι στις γειτονικές χώρες και η προσπάθειά της να επικρατήσουν και να επηρεάσουν τις άλλες περιοχές, τις άλλες χώρες η εξέλιξη ενός παραγωγικού κλίματος ε, παρεμποδίζεται καθώς και η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ και η αποτυχία κατανόησης ε, της ευρωπαϊκής προοπτικής ε, από τους πολιτικούς ηγέτες μετά την διάλυση της Γιουγκοσλαβίας έχει προκαλέσει πολλά αναπάντητα ερωτήματα και εντάσεις σε περιφερειακό επίπεδο και εξακολουθούν να πιστεύει ο κόσμος ε, στο Βολιγράδι ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η κατάσταση. Η Βοσνία απειλείται επίσημα γιατί το Βολιγράδι υποστηρίζει όχι μόνο το status quo αλλά και τις αποσχεστικές τάσεις των Σέρβων ηγετών. Η Σερβία είναι επίσης η μοναδική χώρα στην περιφέρεια που ακόμα δεν έχει αποφασίσει για το μέλλον της. Αν το μέλλον της είναι στην Ευρώπη ή στην επωνομαζόμενη Ανατολή. Η Σερβία είναι ακόμα ε, στο ενδιάμεσο. Να σας ε, πω κάτι που μας ανησυχεί ε, ιδιαίτερα. Μας λένε ότι υπάρχει ανελικρίνεια στην πολιτική της Σερβίας και σε ό,τι αφορά το ιστορικό των χωρών. Παρά κάποιες πρόοδους που έχουν γίνει στη συνεργασία με τις δικαστικές αρχές. Οι πρόσφατες εξελίξεις μας ανησυχούν ιδιαίτερα. Το Βελιγράδι ε, εξακολουθεί να ερμηνεύει την ιστορία του πολέμου με το δικό τους τρόπο. Η δεύτερη εξέλιξη έχει να κάνει μία με την ε, μελλοντική απογραφή που θα γίνει στη Σερβία. που θα περιλάβει και την ε, διασπορά των Σέρβων. Το Μαυροβούνιο εξακολουθεί να θεωρείται μια προσωρινή οντότητα. Γενικά υπάρχουν ανησυχίες ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση υπήρξε αρνητικός αντίκτυπος από την διεθνή οικονομική κρίση. όλα αυτά τα ιστορικά προβλήματα σε όλες τις χώρες και η πολιτική του Βελιγραδίου είναι οι τα βασικά εμπόδια της περιοχής. Ναι, πολλά έχουν αλλάξει χάρη στις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της πολιτικής αιρεσιμότητας, αλλά τα Δυτικά Βαλκάνια δεν έχουν ακόμα εκπληρώσει το δυναμικό τους. Γιατί υπάρχουν ε, ανεύθυνες πολιτικές και ε, εξακολουθεί να υπάρχει διαφθορά. Είναι όλο και πιο σαφές ότι δεν υπάρχει ικανότητα, πολιτική θέληση, πολιτική υπευθυνότητα, πολιτική κουλτούρα για να εφαρμοστεί η ευρωπαϊκή ατζέντα και τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ως εκ τούτου θεωρώ ότι χρειάζεται να δώσουμε μια νέα προσέγγιση προς την περιοχή και να γίνουν πολύ πιο έμεσες και επικοδομητικές προσπάθειες από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταλαβαίνω ότι όλα αυτά είναι πολύ εύκολα να τα πούμε, αλλά πιο δύσκολα να τα πράξουμε. Αλλά θεωρώ και είμαι πεπισμένη ότι ο μοναδικός τρόπος να αντιστρέψουμε την τρέχουσα τάση είναι όλες οι χώρες της περιοχής να λάβουν με καθεστώς υποψήφιας χώρας. Η ρεσιμότητα θα πρέπει να είναι κυρίως κατά αυτών που παρεμποδίζουν τις μεταρρυθμίσεις σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Και η ένταξη στο ΝΑΤΟ σε ό,τι αφορά τη Βοσνία, και τη Μακεδονία είναι απαραίτητη για να βελτιωθεί η ασφάλεια και να επιληθούν ζητήματα στην περιοχή. Κλείνοντας και λαμβάνοντας υπόψη και τα θέματα των ομάδων εργασίας, θα ήθελα να πω ότι οι πολιτικές ατζέντε των κυβερνήσεων της περιοχής δεν είναι απαραίτητα οι ίδιες. Στα Δυτικά Βαλκάνια ποιος πολλής κόσμος ε, θέλει να πάρει χώρα του καθεστώς ε, υποψήφιας χώρας. Δεν είναι μόνο θέμα των ταμείων, των κονδυλίων για την πρωταξιακή φάση παρά το ότι είναι πολύ σημαντικές ε, αυτές οι, αυτά τα κονδύλια. Θα πρέπει όμως να αναλευθούν όλες οι ευθύνες προκειμένου να αποτραπεί ο κοινωνικός ε, η, κοινωνική, ο κοινωνικός ρικοσπαστικός χαρακτήρας. Θα πρέπει να προσεγγίσουμε τους πολίτες στην ε, περιοχή. Αυτό δεν είναι απλό, γιατί μεταξύ άλλων η Ευρώπη θα πρέπει να επιμείνει το κράτος δικαίου, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του πλουραλισμού να κατοχυρωθούν σε αυτές τις κοινωνίες και τέλος είναι πάρα πολύ σημαντικό τα Βαλκάνια να ξεκινήσουν να αισθάνονται ότι ανήκουν στη μία και μοναδική ευρωπαϊκή οικογένεια και ότι μέσα στο πλαίσιο της οικογένειας αυτής η περιφέρεια και οι πολίτες μπορούν να βρουν τις καλύτερες δυνατές λύσεις προς το συμφέρον τους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία μου για την παρουσίασή σας. Να επαναλάβω ότι οι βουλευτές οι οποίοι θα ήθελαν να πάρουν το λόγο στη συζήτηση να συμπληρώσουν παρακαλώ το σχετικό έντυπο. Να συμπληρώσετε το σχετικό έντυπο και να ζητήσετε χρόνο αγόρευσης κατά την Ολομέλεια της 13ης Απριλίου. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να βάλετε και το όνομά σας. Τρία λεπτά για κάθε παρέμβαση. Αν θέλετε να θέσετε μπλε κάρτα, προτιμώ να το κάνετε για τους ομιλητές που είναι στον κατάλογο αγόρευσης. Γιατί όλες οι ερωτήσεις που θα τεθούν στους βασικούς ομιλητές θα απαντηθούν στο τέλος. Στο τέλος λοιπόν, αν θέλετε να κάνετε ερωτήσεις. Να δώσουμε λοιπόν τώρα το λόγο, μάλλον να ξεκινήσει η συζήτηση. Καταρχάς να ακούσουμε τους εκπροσώπους του Αυστριακού Bundesrat. Κύριος Στέφαν Σέναντ, έχετε το λόγο. Άξιο ότι είμαι πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για το λόγο που μου δίνετε. Είναι μια όμορφη ένδειξη και είναι τυχαίο ότι ένας αντιπρόσωπος της Αυστρίας ε, έχει το προνόμιο να ξεκινήσει αυτή τη συζήτηση μετά την ε, ιστορία των Βυτικών Βαλκανίων η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ε, ιστορία της Αυστρίας και της Ουγγαρίας. Γιατί λέμε ότι στα Αυστριακά ότι τα Δυτικά Βαλκάνια ξεκινάνε από τη Βιέννη και αυτό είναι καλό. Στην ε, Ευρώπη, η Ευρώπη χωρίς τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων είναι όπως ένα σπίτι χωρίς στέγη. Τα Δυτικά Βαλκάνια είναι πολύ ιδιαίτερη περιοχή για την Ευρώπη αν θέλουμε να πετύχει η δικαιοσύνη και η ειρήνη η ελευθερία στην ε, Ευρώπη. Θα πρέπει να πετύχει η ενσωμάτωση των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων όσο ε, διαφορετικά και αν είναι τα προβλήματα, όσο και αν είναι δύσκολη η αφετηρία μας, το σημείο αφετηρίας μας. Και φυσικά υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη η κρατική δομή για τη Βοσνία, το πρόβλημα της ε, ασφάλειας στο κοσυφοπέδιο. Αλλά αυτό που είπε η εκπρόσωπος από το Ελσίνκι θα ήθελα να το τονίσω. Έχω ταξιδέψει πολλές στις χώρες των μετικών Βαλκανίων. Η η διαφορά είναι έντονη μεταξύ αυτού που, αυτού που θέλει ο λαός και αυτού που θέλουν οι πολιτικοί ηγέτες. Ιδιαίτερα στο Βελιγράδι μας κάνει εντύπωση αυτό. Γιατί ο κόσμος στο, στην, στο Βελιγράδι λέει «Άμα θέλει να φύγει το κοσυφοπέδιο, ας φύγει». Δεν καταλαβαίνουν γιατί υπάρχει αυτή η αιμονία από τους πολιτικούς ηγέτες. Επίσης η νεολαία χρειάζεται μια προοπτική των Βυτικών Βαλκανίων η νεολαία των Δυτικών Βαλκανίων. Για να μην πέσει στα νύχια του εθνικισμού. Γιατί ο εθνικισμός έχει καταστρέψει πάρα πολλά επί αιώνες στις περιοχές αυτές. Και κατά τους αψούργους έχει τονιστεί και έχει υπεράσει μια άσχημη εικόνα της περιοχής. Θέλουμε λοιπόν μια προπτοκή και είμαι πραγματικά ευγνώμων που επιτέλους ελήφθησε η, απόφαση για τις θεωρήσεις. Γιατί ήταν πραγματικά παράλογο να λένε οι παππούδες στα εγγόνια τι ωραία που ήταν στην εποχή του Τίτο που μπορούσαμε να ταξιδεύουμε που θέλουμε χωρίς ε, θεωρήσεις. Να σκεφτούμε λοιπόν τους νέους. Αλλά φυσικά χρειαζόμαστε και ασφάλεια δικαίου. Φυσικά χρειαζόμαστε προστασία κατά του οργανωμένου εγκλήματος και ε, ενεργή δράση κατά της ε, εγκληματικότητας. Γιατί πρόκειται και για μια περιοχή όπου συχνά ε, υπάρχει εμπορία γυναικών. Και χρειαζόμαστε επίσης και να αντισφαλιστούν τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Και αυτό που χρειάζονται και όλες οι περιοχές και είναι δύσκολο ιστορικά, είναι η συμφιλίωση. Η συμφιλίωση και μία εξίσωση. Και γι' αυτό ευχαριστώ τον Ούγκρο Πρόεδρο και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ανέλαβαν αυτή την πρωτοβουλία μία έκκληση να μην λέμε ότι όλες οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων θα πρέπει να περιμένουν μία την άλλη για να έχουν μία μόνο ε, προοπτική προσχώρησης. Όχι. Μπορεί να είναι διαφορετικά τα πράγματα. Ειδικά για την Μακεδονία, ειδικά για το Μαυροβούνιο, ειδικά για την Αλβανία μπορεί να είναι διαφορετικές οι εξελίξεις. Μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές ταχύτητες στην προσχώρηση. Αλλά τα πράγματα είναι αισιόδοξα. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας. Και τώρα, λέει ο Πρόεδρος, επιτρέψτε μου να σας πω κάτι επιπλέον ενημερωτικά, ότι ο χρόνο αγόρευσης πρόκειται να εμφανίζεται σε αυτήν την ε, οθόνη στα δεξιά μου και έτσι θα ξέρει ο ο μιλητή πόσο χρόνο έχει. επόμενος είναι ε, από την ε, Βρετανική Άνω ο Lord Bones. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βέβαια, ευχαριστώ πάρα πολύ και την Ουγγρική Προεδρία διότι διοργανώσατε αυτήν την σημερινή εκδήλωση για ένα θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ σωστά στην αρχή της ε, ομιλίας μας ε, είπατε το πόσο έχει δεσμευτεί η Ευρώπη ε, όσον αφορά την προσέγγιση της Ευρώπης προς τα Βαλκάνια και αντιστρόφως η πόρτα είναι και παραμένει ανοιχτή όμως παρόλα αυτά νομίζω τώρα θα πρέπει να λαδώσουμε λίγο ε, τους αρμούς της πόρτας διότι ακούγονται κάποιοι τριγμοί στην περιοχή και θεωρώ ότι πρόκειται για μια προτεραιότητα η προτεραιότητα η οποία όμως κατά κάποιο τρόπο έχει α, χάσει κάποιες θέσεις στη λίστα των προτεραιοτήτων οπότε θα πρέπει όλα αυτά να τα προτάξουμε ή στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και και θα πρέπει να είναι κάτι που πρέπει να μας αποσχολήσει ε, περισσότερο. Ε, καταλαβαίνουμε τα οικονομικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε, όμως θα πρέπει να πιεστούν οι κυβερνήσεις ώστε να ανανεώσουμε τις προσπαθίες μας προς εκείνη την κατεύθυνση διότι δεν θα πρέπει οι φίλοι στα δύο Βαλκάνια να θεωρήσουν ότι έχει πέσει το ενδιαφέρον μας για αυτούς και θα έχει σοβαρές συνέπειες κάτι τέτοιο. Πάντως βέβαια είναι ότι δεν μπορεί να τα κάνει όλα και παντού η Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως ούτε εκεί μπορεί να, να, να, να, να θαυματουργήσει η Ένωση, όμως θα πρέπει να θέσουμε κάποιες προτεραιότητες, κάτι το οποίο πάντοτε είναι σωστό. Εγώ κατά τη γνώμη μου σας έχω να προτείνω τα εξής τρία, ότι θα πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στην περιοχή εκείνου, τόσο ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι χώρες θα μπορέσουν να επιβάλλουν ε, το ένα κράτος δικαίου θα πρέπει να αντιμετωπίσουν το οργανωμένο έγκλημα και επομένω είπαμε δεν είναι δυνατό να γίνουν ταυτόχρονα όλα παντού. Άρα να βάλουμε προτεραιότητες στην περιοχή και να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας ή αυτές προς να καταβάλουμε περισσότερες προσπάθειες για να βοηθήσουμε την Βοσνία Ζεγοβίνη και επίσης επίση την προσοχή σας σε ένα άρθρο που εμφανίστηκε χθε από έναν ε, παλαιό συνάδελφό μου στην Άνω Βουλή στην Αγγλία, τον Λόρδο Ashdown που έλεγε ότι αν δεν καταβάλουμε πολλέ προσπάθειε, τότε θα έχουμε γυρίσματα. Κάτι άλλο τώρα γιατί είναι ένα θέμα πάρα πάρα πολύ ευαίσθητο το ότι δυστυχώς ακόμα δεν έχει εξευρεθεί μια λύση όσον αφορά το όνομα, την ονομασία της πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία τη Μακεδονία. Ξέρω ότι εδώ δεν είναι το σωστό φόρο να το συζητήσουμε. Δεν θέλω να κατηγορήσω ούτε τους μεν ούτε τους δε. Εάν όμως στην Ευρώπη το 2011 εάν έχουμε 26 δημοκρατίες που δεν είναι δυνατόν να βοηθήσουν την 27η δημοκρατία, αλλά και άλλη μία δημοκρατία, μία υποψηφία δημοκρατία για να γίνει πλήρες μέλος, τόσο να εξευρεθεί μία λύση, ε, τότε ε, πώς είναι δυνατόν να, να, στρώσουμε το δρόμο για τη διαδρομή που θα κάνει αυτή η χώρα προς εμάς. Επομένως δεν θέλουμε απλώς μία πιο διευρύνη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θέλουμε να μπορέσουμε να χαράξουμε μία κοινή εξωτερική πολιτική. Άρα τέτοιε λύσεις θα πρέπει να αποτελούν προτεραιότητες μας και ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο Πρόεδρος. Εμείς ευχαριστούμε αγαπητέ συνάδελφε και συγχαρητήρια γιατί τηρήσατε ε, με τρομερή ακρίβεια το χρόνο που είχατε, κάτι το οποίο δεν γίνεται κάθε μέρα. Ε, Επόμενος, ε, για τους Πρασίνους. Ουλρίκε Λούνατσεκ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ουγγρική Προεδρία όπως και οι προλαλήσαντε, διότι ανέδειξαν το θέμα των Δυτικών Βαλκανίων σε προτεραιότητα της Προεδρίας και θεωρώ ότι στερούσαμε στο παρελθόν σε σχέση με αυτό, δηλαδή αυτό το όραμα της Θεσσαλονίκης το 2003 πρέπει να παραμείνει ζωντανό. Ε, ξέρουμε ότι υπάρχει μια κόπος λόγω διεύρυνση σε κάποια κράτη-μέλη και το εκτιμούμε όλους ιδιαίτερε που η Ουγγρική Προεδρία το ανέδειξε σε προτεραιότητα. Θα ήθελα να εστιάσω την προσοχή μου σε μία χώρα. Είμαι η συγγήτρια για αυτή τη χώρα ε, στο Κοινοβούλιο. Πρόκειται για το Κωσυφοπαίδιο. Για διάφορου λόγου θα ήθελα να σχολιάσω αυτή. Όπω η Σόνια Πιτσέκ ε, είπε, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, όχι μόνο για το Κωσυφοπέδιο, αλλά για όλες τις χώρες, ότι τα Δυτικά Βαλκάνια ανήκουν ε, στην ενιαία ευρωπαϊκή οικογένεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπόν, ε, θεωρώ, πρέπει να αποστασιοποιηθεί από αυτή την κόπωση που παρατηρείται σε κάποια κράτη-μέλη ως προς τη διεύρυνση και να ε, ε παραδώσετε υπεσχημένα. Σε κάποια κράτη-μέλη ε, υπάρχει με μεγάλη βούληση να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία διεύρυνσης ε, και η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Θα ήθελα λοιπόν να απευθύνω ένα μήνυμα προς τους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Το θέμα των θεωρήσεων για το κοσφοπέδιο. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι όλοι οι υπόλοιποι υπήκοοι των λοιπόν ε, χωρών των Δυτικών Βαλκανίων μπορούν να ταξιδεύουν ελεύθερα για τρίμηνη περίοδο σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός από το κοσφοπέδιο. Και ξέρετε ότι στο Κωσυφοπέδιο υπάρχουν μεγαλύτεροι οπαδοί, μεγαλύτεροι θεασότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ξέρω ότι οι πέντε κράτη-μέλη δεν έχουν αναγνωρίσει ε, το κράτος και υπάρχει ε, ως εκ τούτου νομικό πρόβλημα. Ε, αλλά Σκεφτείτε αυτούς που έβλεπαν μέχρι το πέρας της πρώην Ιουκοσλαβίας ε, να βλέπουν τους γονείς, τους παππούδες να ταξιδεύουν ελεύθερα και εκείνοι οι νέοι τώρα δεν έχουν το δικαίωμα να φύγουν από τη χώρα τους. Δεν έχει σημασία που είναι μικρή η χώρα. Μα φανταστείτε, ε, που, ε, εμάς τους ίδιους ε, βγαίνουμε από το σπίτι μας και πάμε, μπαίνουμε στο αυτοκίνητό μας, στο τρένο, στο αεροπλάνο και πάμε να συναντήσουμε κάποιους. Ε, καταλάβετε ότι ε, κάποιοι δεν έχουν αυτό το δικαίωμα και προς το παρόν η Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Ένωση χάνει την υποστήριξη ε, που είχε στο κοσυφοπέδιο; Δεν είναι τα βλέπω όλα ρόδινα, αλλά απλώς ε, αποτείνομαι στους συναδέλφους που είναι στις, κοινο... που ε, ε, είναι στις κοινοβουλευτικές επιτροπές για τις εσωτερικές υποθέσεις. Παρακαλώ, πιέστε τις κυβερνήσεις σας για να αρχίσει ο διάλογος για τη διευκόλυνση των θεωρήσεων. Η ελευθερία της μετακίνησης και η ασφάλεια είναι οι δύο παράγοντες που καθιστούν απαραίτητη την απελευθέρωση του συστήματος χορήγησης θεωρήσεων. Δηλαδή, ζητάμε από το κοσυφοπαίδιο να έχει καλή τεκμηρίωση, να ακολουθεί τη διαδικασία, αλλά και εμείς πρέπει να κάνουμε ένα ε, βήμα. Σας ευχαριστούμε κυρία μου. Ο κύριος Βόλφαν Γκέρσπρουκ ε, από το Εθνικό Συμβουλίο της Αυστρίας. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, το θέμα το οποίο ε, μας απασχολεί σε αυτή την ε, μεικτή κοινοβουλευτική συνεδρίαση είναι τα Δυτικά Βαλκάνια προς μια καλύτερη ενσωμάτωση και θεωρώ ότι αυτό αποτελεί απόδειξη ότι αυτό είναι η επιθυμία όλων των ε, συμμεταχόντων. Αυτό προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να φροντίσουμε τα Δυτικά Βαλκάνια γρήγορα ή αργά να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους και να καταστούν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ξεκινήσει ως ειρηνευτικό σχέδιο και η Ευρωπαϊκή Ενωπίωση. Και είμαι πεπισμένος ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αν λοιπόν είναι τόσο σημαντικό, θα πρέπει και τα Δυτικά Βαλκάνια προς το συμφέρον μας να καταστούν μέλη. Αγαπητοί συνάδελφοι, να μην κάνουμε το εξή λάθος που έχουμε πολλές φορές κάνει. Να κοιτάξουμε τα Δυτικά Βαλκάνια σαν ανακριτές, σαν δάσκαλοι και να λέμε στους πολιτικούς και στον κόσμο τι να κάνουν. Νομίζω ότι η καλύτερη πρόσβαση είναι να δίνουμε τις ε, συμβουλές μας, να μοιραζόμαστε τις εμπειρίες μας και να τους συνοδεύσουμε σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή από το αυταρχικό κράτος σε ένα δημοκρατικό κράτος. Ε, να αναφερθώ σύντομα στην Αλβανία. Το 2009 είχα την τιμή στα πλαίσια ε, μάλλον της ιδιότητάς μου στα πλαίσια του ΩΣΑ να βρεθώ εκεί και να προβώ σε μία δήλωση μαζί με διάφορους άλλους πολύ έμπειρους συναδέλφους. Ήμουνα στην ε, αποστολή παρατήρησης των εκλογών. Υπήρχαν ε, λάθη αλλά σε γενικές γραμμές εκπληρώθηκαν οι απαιτήσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφέρεται ως παράδειγμα η Αλβανία του αγώνα μεταξύ αντιπολίτευσης και κυβέρνησης. Να αναφέρουμε, το τονίζω αυτό, ότι μια δημοκρατία ε, σημαίνει ότι πρέπει να αποδεχόμαστε το εκλογικό αποτέλεσμα και δεν μπορεί να κρατιέται σε ομοιρία μια χώρα α, από αυτούς που δεν αποδέχονται το εκλογικό αποτέλεσμα, ακόμα και αν είναι δημοκρατικές δυνάμεις. Νομίζω ότι το οφείλουμε σε όλες τις χώρες, όχι μόνο στην Αλβανία, να είμαστε αντικειμενικοί. Και όχι να ορίζουμε από τράγου, τράγους, να τους βοηθήσουμε σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή που έχουν να διανύσουν τα ευρωπαϊκά κράτη χρειάστηκαν 100 χρόνια παραπάνω για να πετύχουν τη δημοκρατία και τους ζητάμε από αυτές τις χώρες να το κάνουν σε κάποια χρόνια, σε κάποιες δεκαετίες. Είναι λογικό ότι υπάρχουν δυσκολίες. Θα πρέπει να τους δώσουμε τον κατάλληλο χρόνο για να υπάρξουν αυτές οι εξελίξεις για τη δημοκρατία. Δεν είναι μόνο θέμα ε, μυαλού αν θέλετε, εγκεφαλικό, είναι θέμα της καρδιάς. Εκεί θα πρέπει να έχει τις ρίζες της η δημοκρατία και θα πρέπει λοιπόν να συνδράμουμε, να συμβάλλουμε να μπορέσουν αυτές οι χώρες ε, να έχουν στην καρδιά τους τη δημοκρατία και θεωρώ ότι όλες οι χώρες των Βαλκανίων ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ε, ζητήσατε μπλε κάρτα. 30 δευτερόλεπτα έχετε στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Μπούζεκ. Θέλω να ρωτήσω τη Σόνια Βίσεκ κάτι. Πολύ ισορροπημένη ήταν η εισαγωγή που έκανε. Με εξέπληξε. Με εξέπληξε η ανάλυση της για τα Δυτικά Βαλκάνια. Κάτι δεν ήταν ακριβές. Είναι το θέμα των θρησκευτικών αποχρώσεων. Υπάρχουν τουλάχιστον δύο χώρες, δύο εκκλησίες που έχουν τεράστια προβλήματα διότι δεν αναγνωρίζονται η Ορθόδοξη Εκκλησία του Μαυροβουνίου από τη μια πλευρά και η Ορθόδοξη Εκκλησία τη Μακεδονία λέει ο μιλητή από την άλλη. Και η Ορθόδοξη Εκκλησία και ο νέο πατριάρχη τη Σερβία ήταν πολύ αποτελεσματικό για την άρση κάποιων εμποδίων στην περίπτωση του Κωσυφοπεδίου. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι τα σχόλιά σα. Υπάρχει κάτι που πρέπει να υποθεί επ' αυτού, επ' αυτή τη ευκαιρία. Και εφόσον έχω το μικρόφωνο, δράτω με τη ευκαιρία να απευθύνω άλλη μια πρόκληση. Υπάρχει ένα πρόβλημα με την ονομασία για τη Μακεδονία, λέει ο μιλητής. Έχω μια πρόταση. Η Μακεδονία μας, Νάσα Μασεντόνια, Our Μασεντόνια, είναι πολύ διαφορετικό από τη Βουλγαρική Μακεδονία και από την Ελληνική Μακεδονία. Ίσως αυτή είναι μια διέξοδος. Να ξεκινήσει ο διάλογος, να βρεθεί μια λύση να δοθεί μια προθεσμία και να επιταχυνθεί η διαδικασία της ε, ολοκλήρωσης στα Δυτικά Βαλκάνια. Ευχαριστώ. Ήταν λίγο περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα, αλλά πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε. Κυρία μου, αν έχετε την καλοσύνη να απαντήσετε αμέσω τώρα. Ευχαριστώ για αυτό το ερώτημα. Δεν είχα εστιαστεί επί θρησκευτικών θεμάτων, αλλά η Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία είναι από τους βασικούς θεσμούς της Σερβίας ιστορικός και τώρα όχι μόνο σαν θρησκευτικό θεσμό αλλά σαν θεσμός που εδράζεται επί της ερβικής ταυτότητας και στον Ορθόδοξο κόσμο οι Ορθόδοξες εκκλησίες είναι εθνικές εκκλησίες και αν δεν αναγνωρίζεται η εκκλησία του Μαυροβουνίου και της Μακεδονίας λέει η ομιλήτρια, ε, είναι σαν να παρνιέται κανείς αυτές τις χώρες και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι ξέρουμε σαφώς ότι η Μακεδονική Εκκλησία λέει ομιλήτρια ταυτίζεται με μακεδονική ταυτότητα λέει και με το μακεδονικό λαό λέει η ομιλήτρια και έχουμε κι άλλο ένα πρόβλημα που αναφύεται. Η μη αναγνώριση της Ρουμανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στη Σερβία. Η Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία θα έπρεπε και θα μπορούσε να διδραματίσει σημαντικό ρόλο αν ο Πατριάρχης συνεχίσει την πολιτική άρσεως των εμποδίων. Για την ώρα το έκανε αυτό μόνο στην περίπτωση Κωσυφοπεδίου. Ελπίζω να κάνει και κάτι και προς τη Μακεδονία, λέει Μιλήτρια, και προς το Μαυροβούνιο. Αυτό ελπίζουμε Ελπίζουμε, δεν ξέρω αν θα γίνει αρκετά σύντομα. Θα ήθελα να τονίσω εκ νέου την ανάγκη που υπάρχει ε, να υποστηριχθεί υποψηφιότητα των χώρο στην περιοχή για να σταματήσουν οι αρνητικές διαδικασίες στην περιοχή και θα τεθεί τέρμα στα προβλήματα τα διάφορα που υπάρχουν. Χρειάζεται η αντίστροφη διαδικασία να ακολουθηθεί, δεν θα είναι εύκολη, θα έχει ανωδικές ή καθοδικές πορείες για κάθε χώρα, χρειάζεται όμως το πλαίσιο για την οικοδόμηση του συστήματος. Σήμερα έχουμε μόνο τους νόμους που ψηφίζονται και ψηφίστηκαν πρόσφατα αλλά δεν εφαρμόζονται. Και κάτι πολύ κρίσιμο είναι να υπάρχει μεγαλύτερη εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών διότι αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι, οι οποίοι πραγματικά είναι ευρωπαϊκές δυνάμεις στη χώρα και θα μπορούσαν να βοηθήσουν να πιεστεί η κυβέρνηση. Μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση σε κάποιο βαθμό κατέβαλε σχετικές προσπάθειες, αλλά όχι πραγματικά, διότι ε, λειτουργεί κυρίως μέσω των κυβερνήσεων. Αυτή η νέα προσέγγιση θα βοηθούσε. Δηλαδή να στραφούμε προ τη βοήθεια των κοινή των πολιτών. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο ότι μπορεί να σηκώσετε μπλε κάρτα για να απευθύνεται ένα ερώτημα σε οποιονδήποτε ομιλητή από τον κατάλογο. Από το Ουγγρικό Κοινοβούλιο, επόμενο ομιλητή. Ο συνάδελφο ο κ. Ρίτσαρτ Χέρτσιγκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Όπω βλέπετε, τους τελευταίους μήνες τα οικονομικά ζητήματα ήταν στο επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Πολιτικού προγράμματο. και θα πρέπει να βρεθεί λύση στην κρίση. Όμως τα οικονομικά προβλήματα δεν θα πρέπει να επισκιάζουν τη διεύρυνση. Πρέπει να παραμείνει ανοιχτή η Ευρωπαϊκή Ένωση προς τις χώρες εκείνες που πληρούν τα κριτήρια ένταξης και είναι έτοιμες να εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις στο πνεύμα των ευρωπαϊκών αρχών. Η Ουγγρική Προεδρία ε, θέλει να συνεχιστεί η διαδικασία των διευρύσεων. Συνεργαζόμαστε λοιπόν γι' αυτό χέρι με χέρι με τα κράτη-μέλη, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις υποψήφιες χώρες, ούτω ώστε να γίνουν βήματα πρόοδου. Κύριε Πρόεδρε, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που ενταξιακέ διαπραγματεύσεις με την Κροατία φτάσαν στο τελευταίο στάδιο. Σημαντική πρόοδος έχει γίνει σε αρκετούς τομείς, όμως ε, πολλές προκλήσεις εξακολουθούν να υπάρχουν στις υποψήφιες χώρες και αυτές που θέλουν να υποβάλουν υποψηφιότητα. Σε κάποιες χώρες της διεύρυνσης η ορμή των μεταρρυθμίσεων πρέπει να στεθεί επί της ορτής διακυβέρνησης, τη βελτίωση του κράτους δικαίου, επιτάχυνση της οικονομικής μεταρρύθμισης και βελτίωση να προσαρμοστούν και να εφαρμόσουν το κεκτημένο. Το κοινοτικό αυτή η πρόοδος αντιμετωπίζει διάφορες δυσκολίες με πιο εστιασμένη τεχνική βοήθεια σε αρχικό στάδιο θα μπορούμε να του βοηθήσουμε. Και η βοήθεια αυτή θα μπορεί να συμβάλλει περισσότερο στι προσπάθειε που καταβάλουν οι χώρε και θα καλυφθούν καλύτερα και ανάγκε του. Από τη στιγμή που θα πληρούνται όλα τα κριτήρια, η ένταξη της Κροατίας θα στείλει θετικό μήνυμα, πιστεύω, θετικό σήμα στα υπόλοιπα Δυτικά Βαλκάνια και θα συμβάλλει έτσι στη σταθερότητα σε όλη την περιοχή. Αυτό το θετικό παράδειγμα της ε, Κροατίας θα παροτρύνει και άλλες χώρες της ε, περιοχής να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για να φτάσουν στις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η υλοποίηση, η πραγματοποίηση πραγματικών μεταρρυθμίσεων οδηγεί σε απτά αποτελέσματα για τους πολίτες. Η Μακεδονία, ο μιλητής, το Μαυροβούνιο και η Σερβία ε, μπήκαν στο καθεστώς απελευθέρωσης από τις θεωρήσεις το 1999. Το ίδιο και για την Αλβανία, Βοσνία και Ζεγοβίνη, ξεκινώντας από το 2010. Οι άλλες μπήκαν το 2009, ζητά συγγνώμη διερμηνέας. Λοιπόν, πρέπει να, αντιστραφεί, να καταπολεμηθεί και η παράνομη μετανάστευση. Αυτό συμβάλλει αυτή η απελευθέρωση. Πρέπει όμως να ισχύσει αυτό καθεστώ για όλα τα Δυτικά Βαλκάνια. Η αδίποτε πρόοδο στον τομέα πρέπει να εδράζεται επί της αξίας των προσπαθειών καταβάλλονται. Η διεύρυνση είναι βασικό οδηγό για οικονομικέ και πολιτικέ μεταρρυθμίσει που ανοίγουν το δρόμο για σταθερότητα και ευμάρεια όλη τη περιοχή. Ευχαριστώ, συνάδελφε. Ε, θα ζητήσω παρέμβαση από πλευρά της κυρίας Doris Πακ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και ο συνάδελφος Γέλκο Κάτσιν σε λίγο, σε τέσσερα λεπτά. Οι κυρίες έχουν πρώτε το λόγο. Ορίστε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, συνάδελφοι. Θα ξέρετε ότι εδώ και 22 χρόνια εργάζομαι για τις χώρες στα Δυτικά Βαλκάνια. Υποφέρω και χαίρομαι μαζί τους, αλλά έχω και απογοητευτεί. Όχι σε όλα, αλλά σε πολλούς τομείς. Υπάρχουν πολλές ε, ε, πολλοί λόγοι για να χαίρομαι, αλλά κοιτάζοντας την Βοσνία Ερσεγοβίνη, το Κωσυφοπέδιο, την Μακεδονία, πρέπει να σας πω ότι κάτι με λυπεί είναι ότι δεν έχει βελτιωθεί η κατάσταση για τον κόσμο. Δεν είναι οι πολιτικοί στη Βοσνία Ερσεγοβίνη αυτοί που αναλαμβάνουν την ευθύνη τους για να ξεπεράσουν τις εθνοτικές διακρίσεις και στη χώρα αυτή υπάρχουν τρεις ε, διαφορετικές ε, εθνότητες και πολλοί που δεν ανήκουν σε καμία από αυτές. Όλοι είναι πολίτες της Βοσνίας Αρζεγοβίνης. Δεν τα ξεκαθαρίζουν όμως οι πολιτικοί αυτά και παίζουν ε, με τις εθνοτικές αυτές μειονότητες. Γι' αυτό θα ήθελα πιο μεγάλες προσπάθειες από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την κατεύθυνση αυτή για να αναγκαστούν οι πολιτικοί να εργαστούν για την ευημερία των πολιτών και όχι μόνο να σκέφτονται τα δικά τους. Να σκεφτούν οι πολιτικοί ότι θα πρέπει να μας απασχολήσουν θέματα εκπαίδευση Ποιο θα επενδύσει στη Βοσνία Ερζεγοβίνη αν δεν υπάρχει κόσμο με την σωστή εξειδίκευση που θα δουλέψει καλά. Έχουμε χάσει πάρα πολλές ευκαιρίες και χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον τελευταίο καιρό έχει δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Για το Πέδιο θα πρέπει να σας πω ότι θα πρέπει να προσέξουμε τις γειτονικέ ε, χώρες. Θα πρέπει να συνεχιστεί ο διάλογος με τη Σερβία, λαμβάνοντας υπόψη όσα χρειάζονται για τη ρύθμιση της ζωής του κόσμου. Μιλάμε για τις ε, όλες τις μειονότητες οι οποίες θα πρέπει να ζουν αρμονικά χωρίς να ενοχλούν το Βελιγράδι. Δεν είναι δυνατόν να θέλει κανείς να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να έχει τόσα προβλήματα με το κοινωνική του χώρας. Και να πω ότι αυτό που υποφέρει η Μακεδονία εδώ και πάνω από μία δεκαετία είναι ντροπή για μας. Δεν είναι δυνατόν ένα ευρωπαϊκό κράτος να εμποδίσει με τέτοιο τρόπο την προσχώρηση της Ευρωπα... στην Ευρωπαϊκή Ένωση τέτοιο τρόπο. Και οι Έλληνες λοιπόν θα πρέπει να αναρωτηθούν. Δεν είδατε ότι υπάρχουν άλλες δυνατότητες και μπορεί να υπάρχει η εγώ είμαι υπέρ τη λύση τη διπλή ονομασία, αλλά δεν είμαι υπέρ του να μην διατηρηθεί ο όρο Μακεδονία, γιατί δεν πρέπει να αφαιρέσουμε την ε, ταυτότητά του. Η Κροατία. Έχουν τεθεί πολύ υψηλοί στόχοι που δεν είχαν τεθεί για τους ε, Βούλγαρους και τους Ρημάνους. Και γι' αυτό αντιμετωπίζουμε τώρα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολύ ψηλά πρότυπα για τους Κροάτες. Δεν θα μιλήσω για τις υπόλοιπες χώρες, δεν θα μιλήσω για την Αλβανία για να μην με μαλώσει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής. Η κυρία Ροδούλα Ζήση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Αν θα μπορούσατε να σηκώνεστε για να μιλήσετε, για να σας βλέπουμε, θα ήταν πολύ πιο εύκολο για μας. Αν θέλετε λοιπόν, κυρία μου, αν θέλετε να σηκωθείτε να σηκωθείτε παρακαλώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί έτσι μπορώ να σας βλέπω. Πολύ καλύτερο αυτό για μένα. Σας ευχαριστώ. Okay, thank you very much. ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε ε, και θέλω να σας συγχαρώ εκ μέρους της ελληνικής αντιπροσωπείας, της κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας, για αυτή την πρωτοβουλία που επιβεβαιώνει τελικά ότι η πολιτική ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δίπολο εμβάθυνσης και διεύρυνσης αποδεικνύει ότι τελικά η ευρωπαϊκή ένωση δεν είναι μια λέσχη δυτικοευρωπαϊκών κρατών αλλά είναι μια αρχή μια συλλογική κοινωνική πολιτική και οικονομική οντότητα που θέλει να ενσωματώσει όλο και περισσότερα μέλη της βάσει όμως των θεμελιωδών αξιών ε, της δημοκρατίας του κράτους δικαίου του σεβασμού των δικαιωμάτων και των ελευθεριών και των φιλικών και ειρηνικών σχέσεων μεταξύ των λαών. η ελλάδα κύριε πρόεδρε είναι από τις χώρες εκείνες όλη η Βουλή, ε, η χώρα μας, οι κυβερνήσεις που έχουν στηρίξει διαχρονικά την ε, είσοδο των Δυτικών Βαλκανίων στις δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα έχουμε πρωτοπορήσει σε αυτό το θέμα γιατί όπως ξέρετε η ατζέντα στην Προεδρία την, Ελληνική της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2003 έλεγε ακριβώς αυτό το στόχο και σηματοδοτούσε αυτό το όραμα της μεγάλης οικογένειας των δυτικών ε, βαλκανίων μέσα στη μεγάλη οικογένεια της ευρωπαϊκής ένωσης. υπάρχουν όμως περιφερειακά προβλήματα υπάρχουν αδυναμίες και πρέπει να το πούμε εδώ ότι έγινε και μια ε, αν μου επιτρέπετε τον όρο έγινε μια κοιλιά σε ό,τι αφορά αυτό το στόχο αυτή τη στόχευση τα προηγούμενα χρόνια. γι' αυτό και πάλι χαιρόμαστε για αυτή την πρωτοβουλία και η ελλάδα επανασηματοδοτεί αυτό τον οδικό χάρτη για, την, ε, το 2014 έτσι ώστε πραγματικά τα δυτικά βαλκάνια να εισέλθουν στην ευρωπαϊκή οικογένεια. επειδή αναφέρθηκαν εδώ κάποια πράγματα πρέπει να πω ότι και για την πρώην ιουγκοσλαβική δημοκρατία της μακεδονίας η χώρα μας στάθηκε αρρωγός και σε δύσκολες στιγμές και υποστήριξε αυτή την ένταξη και βοήθησε η χώρα μας και ε, με, το σχέδιο ανασυγκρότησης της περιοχής. Όμως δεν πρέπει να υπάρχουν παρερμηνίες στις ιδιαίτερες περιφερειακές ιστορικές ανάγκες, συνεργασίες, συμφωνίες. Διότι πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρα ότι προκειμένου η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ληφθούν και από την ευρωπαϊκή ένωση όλες αυτές οι ιδιαιτερότητες της περιφέρειας. κοινή αποδεκτή λύση στο ζήτημα της ονομασίας λύση που θα έχει γεωγραφικό προσδιορισμό έναντι όλων. εμείς ε, πιστεύουμε ότι αυτή η περίοδος που δεν βοήθησε για να προχωρήσουμε σε αυτό το όραμα αφορούσε στην οικονομική κρίση αφορούσε στα θέματα εμβάθυνσης αλλά τώρα είναι η ώρα και συμβάλλουμε κι εμείς προς αυτή την κατεύθυνση αξίζει να τονίσουμε τελικά ότι υπάρχουν ζητήματα που έχουν να κάνουν με αυτά που θα συζητήσουμε πιθανώς στα working groups ζητήματα δικαιοσύνης και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν ζητήματα διαφθοράς και οργανωμένου εγκλήματος υπάρχουν τα προβλήματα της μετανάστευσης της παράνομης το human trafficking υπάρχουν θέματα με τα ανθρώπινα δικαιώματα. πιστεύω κύριε πρόεδρε πιστεύω αγαπητοί και αγαπητές ε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι ότι χρειάζεται η ευρώπη να αποδείξει ότι μπορεί και όλοι μαζί σεβόμενοι τις αρχές του δικαίου να προχωρήσει στη διεύρυνση ενσωματώνοντας τα δυτικά βαλκάνια. η πολιτική της διεύρυνσης είναι αναμφισβήτητα η πιο πετυχημένη έκφραση της κοινή εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας. ενοποιούμε την ήπειρο και πετυχαίνουμε να επεκταθεί η ζώνη ασφάλειας η ζώνη συνεργασίας η ζώνη καλής γειτονίας και στις περιφερειακές περιοχές ε, και περιφερειακές συνεργασίες. Έχουμε ανάγκη από όρομα, έχουμε ανάγκη από στόχους, έχουμε ανάγκη να συμβάλλουμε όλοι, όχι απλά τεχνοκρατικά και με λίγο πάθος, με λίγη καρδιά και γνώση της ιστορίας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος, για την παρέμβασή σας. Ο επόμενος ομιλητής προέρχεται από την ε, Λιθουανία. Ο κύριος Κάιντες. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ διότι μας δίνετε την ευκαιρία να εκπροσωπήσουμε τη χώρα μας. Είχα την ευκαιρία, ξέρετε, επανειλημμένα να επισκεφθώ τα Δυτικά Βαλκάνια και έγινα μάρτης των πρόοδων που έχουν σημειωθεί. Στις 28 ε, του Μαρτίου ο Γιώσεπ ε, επισκέφθηκε τη χώρα μας. Επίσης, στην χώρα μας ήρθαν και άλλοι εκπρόσωποι, εκπρόσωποι της χώρας του Μαυροβουνίου, της Βοσνίας Ατζεκοβίνης. Η χώρα μας, ξέρετε, έχει στενές σχέσεις με τις χώρες εκείνες. Ξέρετε, ε, μας αρέσει το μπάσκετ. Και οπότε καταλαβαίνετε, επίση ε, έχουμε αναπτύξει και οικονομικέ και εμπορικέ σχέσει, όμω από την άλλη μεριά τα παράπονά μα είναι το επίπεδο τη διαφθορά. Έχουμε επομένω ένα σωρό προβλήματα που θα πρέπει σιγά σιγά να δούμε πώ θα επιληθούν και πιστεύουμε ότι η Κροατία θα μπορέσει τον Ιούλιο φέτο να ολοκληρώσει τι διαπραγματεύσει τη προσχωρήσεω. Την ε, τα τέλη του έτου, κατά φθινόπωρο, πρόκειται να προχωρήσουμε περαιτέρω. Το ίδιο συμβαίνει για το πέδιο. Τώρα από την άλλη μεριά Φιρόμ, Ελλάδα έχουν περιπλέξει τα πράγματα και νομίζω ότι θα πρέπει να βοηθήσουν κάπως ε, οι, τις Ευρωπαϊκές Η Βοσνία Ζεγοβίνη απαιτεί να ασχοληθεί περισσότερο μαζί της η Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο νομίζω θα ήταν χρήσιμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρετε, τώρα ε, πάσχει, πάσχει από αυτήν την κόποση της ε, διεύρυνσης και δεν μπορούμε παρά να διαπιστώσουμε ότι περαιτέρω διευρύνσεις έτσι εμποδίζονται. Και επομένω αυτό το οποίο θα ήταν θετικό θα ήταν οι νέοι στα Δυτικά Βαλκάνια να μπορούν να διακινούνται, να ταξιδεύουν, να κυκλοφορούν ευκολότερα στην Δυτική Ευρώπη. Νομίζω αυτό θα ήταν ένα βήμα πρόοδου. Έτσι θα είχαμε καλύτερε σχέσει. Ο πρόεδρο. Α, πολύ ωραία. Βλέπω και μία μπλε γαλάζια κάρτα κάπου υψώθηκε. Ποιο την εσήκωσε την κάρτα. Μήπω και εσεί, ο κύριο Αντριοκάτη, και εσεί είχατε σηκώσει, θέλετε επίση και μία ερώτηση. Είχατε ερώτηση. Μπορείτε μετά την αγόρευση να προσθέσετε την ερώτηση. Αντριουκάιτε. Ναι, έχω μία ερώτηση, λέει ψώντα την γαλάζια κάρτα. Η ερώτησή μου, ξέρετε, απευθύνεται εις ε, τον ε, πρόεδρο ή την πρόεδρο της ε, Κροατικής Βουλής. Τον κύριο, τον κύριο Μπέμπιτς. Τι έχετε να πείτε για αυτό το δημοψήφισμα που θα κάνετε το φθινόπωρο. Ποια ημερομηνία θα γίνει το δημοψήφισμα και πέστε μας αν προσδοκάτε κάποια θετική ε, απάντηση σε αυτό το δημοψήφισμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτησή σας. Αν λήξουν οι διαπραγματεύσεις μέχρι το τέλος Ιουνίου, όπως δηλαδή το έχουμε σχεδιάσει. Μετά το ψήφισμα του Κοινοβουλίου, λοιπόν, μπορεί να γίνει το δημοψήφισμα για να υπογραφεί η συμφωνία. Δηλαδή είμαστε έτοιμοι. Μπορεί να διεξαχθεί σε αρχές φθινοπόρου το δημοψήφισμα. Αν περατωθούν οι διαπραγματεύσεις μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Εάν όχι, γιατί μην ξεχνάτε ότι έχουμε και εκλογές ε, στην ε, Κροατία, ε, τότε δεν θα μπορέσει να διεξαχθεί το δημοψήφισμα το φθινόπωρο. Δηλαδή είναι δύσκολο να οργανώσουμε εκλογές και δημοψήφισμα ταυτόχρονα. Θα δούμε αν μπορούμε τελικά να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα. Μπορεί να γίνει πρώτα το δημοψήφισμα και μετά ε, να διεξαχθούν οι εκλογές για να μην τις βαρύνουμε με ευρωπαϊκά ζητήματα, να εστιάσουμε στα εθνικά μας ε, θέματα. Υπάρχει πάντως διακομματική συνένεση και για την αμυντική πολιτική, για την εξωτερική πολιτική, την προσχώρηση στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλό θα ήταν να διαχωρίσουμε τα εθνικά από τα ευρωπαϊκά θέματα. Ε, έχουμε σημειώσει καθυστέρηση αληθεύει αυτό. Οι πιο ευρωσκεπτικιστές θα γίνουν πιο πολύ άριθμοι αν καθυστερήσουμε και άλλο. Δεν νομίζω όμως ε, να τεθεί υπό αμφισβήτηση η προσχώρηση της Κροατίας στην Ένωση. Ελπίζω να μην είναι αρνητική έκβαση του δημοψηφίσματος. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο Πρόεδρος ε, ε, του Ουγγρικού Κοινοβουλίου θα αναλάβει τώρα την ε, Προεδρία. Ευχαριστώ. Έχετε το λόγο. Κύριε Μπούζεκ, αγαπητέ Πρόεδρε του Ουγγρικού Κοινοβουλίου, σας ευχαριστώ και τους δύο για την ε, συνδιοργάνωση της σημερινή συζήτησης που έχει ιδιαίτερη σημασία και για τα θεσμικά μας όργανα αλλά και κυρίως για τους λαούς των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Κύριε Μπίμπιτς, ε, θα αρχίσω την ομιλία μου ευχαριστώντα σας ε, για τα όσα έχετε κάνει για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Ένα βασικό πρόβλημα στα Δυτικά Βαλκάνια είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς και της ε, οργανωμένης εγκληματικότητας. Ναι οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων συνεργάζονται και εκδίδουν μεταξύ αυτών τους ε, ε, εγκληματίες. Αυτό είναι καλές οι χώρες, αλλά στην καταπολέμηση της διαφθοράς δεν τα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Εκτός από τον καλό του μαθήτη την Κροατία, που έχει πολύ καλές επιδόσεις και νομίζω ότι πρέπει να αποδώσουμε τα εύσημα στη χώρα για τις προσπάθειές της. Ε, σας συγχαίρω παρότι δεν είμαστε από την ίδια πολιτική οικογένεια. Οφείλω να αναγνωρίσω τα, τα επιτέγματά σας ε, στις προσπάθειες που κάνετε για την εξάλληψη της διαφθοράς. Ε, θα ήθελα τώρα ε, να ε, σχολιάσω αυτές τις επιταγές εν λευκό που δίνουμε στα μέλη του Σερβικού Κοινοβουλίου. Δεν το καταλαβαίνουμε ακριβώς γιατί συμβαίνει αυτό. Θα θέλαμε οι συνάδελφοι από τη Σερβία να λάβουν υπόψη τις συστάσεις του Συμβουλίου της Βενετίας για να δοθεί ε, μία λύση στο πρόβλημα της Σερβίας, διότι πλήττεται ε, η ίδια η αξιοπιστία της χώρας. Ελπίζουμε ότι θα ρυθμιστεί το πρόβλημα το ταχύτερο δυνατόν. Ε, κλείνοντας να πω και κάτι άλλο για την ε, Σερβία. Ο κυρία Λουνατσέκ είπε ότι είχαν έρθει τρεις ε, δήμαρχοι από το Κωσυφοπέδιο και από κάποιες σερβικές ε, δημοτικές αρχές. Όλοι αυτοί που ήρθαν ήταν φιλελεύθερου προσανατολισμού, α το θέσω έτσι. Τέλο πάντων, το σημαντικό είναι που είναι ανοιχτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για όλε τι αυτοδιοικητικέ αρχέ. Νομίζω, Πρόεδρε, ότι πρέπει να ανταμείβονται όσοι βρίσκουν ταχύτατα λύσει στα προβλήματα και πρέπει να αναγνωριστεί το πόσο ε, γρήγορα ε, ρυθμίστηκε η θεσμική κρίση στο Κωσυφοπέδιο. Εξελέγει νέο Πρόεδρο. Δεν θα ήταν σωστό να προσκαλέσετε και τον νέο Πρόεδρο στο Κοινοβούλιο για να δούμε νέα πρόσωπα και έτσι να υιοθετήσουμε ίσως και μια ε, ανανεωμένη προσέγγιση, μια νέα προοπτική. Ε, να δώσουμε, να τονώσουμε την, ε, το διάλογο που ίσως έχει επέλθει σε τέλμα. Μπορούσατε στη διάσκεψη των Προέδρων παρακαλώ να το θέσετε το θέμα. Κύριε Βούζεκ, να προσκαλέσετε τον Πρόεδρο. Ευχαριστώ. Ο επόμενος. Ο επόμενος, λοιπόν, από το Ηνωμένο Βασίλειο. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Είναι μια καλή διάσκεψη αυτή που πραγματοποιείται επί Ουγγρικής Προεδρίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα για το μέλλον της Ευρώπης. Από την έποψη του Ηνωμένου Βασιλείου πρέπει να πούμε ότι όλα τα πιο βασικά κόμματα της, του Ηνωμένου Βασιλείου είναι υπέρ της συνεχιζόμενης διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και θεωρείται σαν ευρωσκεπτιστική χώρα πολύ συχνά η Βρετανία, αλλά παραδέχεται η Βρετανία πολύ συχνά ότι μέσω της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ενώσεως η σταθερότητα και η ειρήνη και η ελευθερία ε, εξαπλώθηκε σε πολύ μεγαλύτερη έκταση της Ευρώπης από ό,τι ήταν δυνατόν διαφορετικά και αυτά τα ωφέλη ε, τα απολάμβανε η Δυτική Ευρώπη επί πολλές δεκαετίες, η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη για μικρότερο χρονικό διάστημα. Εμείς χρωστάμε στα Βαλκάνια να τους δώσουμε τη δυνατότητα αν θέλουν και εκείνα να αποκτήσουν αυτά τα αγαθά, να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να ωφεληθούν από την ειρήνη, σταθερότητα, ε, ανθρώπινα δικαιώματα, κράτος δικαίου και όλα τα κριτήρια της Κοπενχάγης που είναι διαθέσιμα σε αυτούς αν τελικά τους αφήσουμε να γίνει αυτό. Στη Βρετανία και σε άλλα μέρη της Ευρώπης τα προσεπήρηση προβλήματα πριν λάβει η χώρα η διεύρυνση είναι εκείνα που ήδη αναφέρθηκαν. Το οργανωμένο έγκλημα, μετανάστευση, μεθοριακός έλεγχος, έλεγχος των συνόρων. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι αυτοί οι τομείς πολιτικής έχουν εξομαλυνθεί, έχουν λυθεί τα προβλήματα για να γίνει ένταξη πρέπει να συνεχιστεί η όθηση προς διεύρυνση και να πραγματοποιηθούν αυτά γρήγορα. Ένας τομέας ο οποίος πιστεύω είναι ξεκάθαρος για τα Δυτικά Βαλκάνια που μας που τα βλέπουμε από μακριά είναι αυτά που ανέφερε η Βοσνία Ζεγοβίνη. Αυτά τα θέματα που αναφέρθηκαν χρειάζουν ιδιαίτερη ειδική προσοχή από την Ευρώπη. Σαν Ήπειρος δεν μπορούμε να δεχτούμε να κινηθεί προς τα πίσω η Βοσνία προς τα προβλήματα του είδους που υπήρχαν δεκαετία του 90 και το δεκαετία του 2000. Όχι στην ίδια κλίμακα να υπάρχουν. Δεν μπορούμε να χάσουμε την επιτευθύσα πρόοδο. Και πιστεύουμε ότι αυτή είναι σημαντική διάσκεψη, γιατί τα εθνικά κοινοβούλια μπορούν να ασκήσουν πιέσει, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ασκήσει πιέσει ούτω ώστε το Συμβούλιο να, να εστιάζεται από αυτών των θεμάτων και να μην εστιάζεται τόσο όσον αφορά την ε, Ένωση της Μεσογείου. Αν σταματήσουμε να ανησυχούμε για αυτά τα θέματα περισσότερο και συνεχίσουμε με την ολοκλήρωση των Δυτικών Βαλκανίων θα είναι κάτι πολύ θετικό. Θα ήθελα η Σόνια Μπζέρκο που η παρουσίασή της ήταν έξοχη ε, αναφέρθηκε σε πολύ εφάνταστο τρόπο για το μέλλον, στο τέλο τη διασκέψεως θα ήθελα να ξέρω ακριβώ ποια μορφή θα μπορούσε να έχει αυτό ο εφάνταστο δρόμος ε, προ τα μπρό. Θέλω να πω ότι μπαίνουμε στη φάση της ύφεση στα Δυτικά Βαλχάνια και στη Βοσνία και... Ε, την το επόμενο φινόπορο μπορεί να κερδίσουν τα προοδευτικά κόμματα. Πρέπει να δοθεί δυνατότητα υποψηφιότητα σε όλους χωρίς να επιμένουμε τόσο επί των κριτηρίων, διότι η υποψηφιότητα είναι μακρά διαδικασία, είναι πιο δημιουργική από αυτή που είμαστε μέσα τώρα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τμήμα της διαδικασίας και η διαχείριση γίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. είναι πιο ελεγχόμενη η εξέλιξη, κυρίως μέσω των θεσμικών οργάνων της επιβολής του νόμου και η προσέγγιση προς την κοινωνία των πολιτών και προς όλα τα εμπλεκόμενα και ενδιαφερόμενα μέρη που ενδιαφέρονται να γίνει ένταξη στην Ευρώπη. Η προσέγγιση πρέπει να είναι πιο δημιουργική, να υπάρχει πρόσβαση για όλους την περιοχή σε αυτές τις διαδικασίες. Διότι παραδείγματος χάρη μπορούμε να αναπτύξουμε μια εκστρατεία προς την κοινωνία των πολιτών για να γνωστοποιηθεί το πρόγραμμα τη Ευρωπαϊκή Ενώση στο ευρύτερο κενό. Να κινητοποιηθούν οι πολίτε, να πιέσουν την κυβέρνηση για να δώσει περισσότερα. Σύμφωνα με τα δικά του σχέδια δράση. Γι' αυτό ζητούμε βοήθεια και την Ευρωπαϊκή Ένωση και από αλλού. Δυστυχώ η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι πολύ ευέλικτη για να ε, ξεκινήσουν αυτή την εκστρατεία. Θέλουμε υποστήριξη από αλλού. Διότι χρειάζεται μια όθηση, μια ορμή για τη Σερβία κυρίως, για να κινητοποιηθούν οι πολίτες, γιατί έχουν απογοητευτεί με την κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν πολύ μεγάλες προσδοκίες και πολύ λίγα αποτελέσματα είδαν. Και αυτό μπορεί να του κάνει να υπομισθούν τι ευθύνε του για το δικό του μέλλον. Πρέπει να καταλάβουν ότι δεν φταίει μόνο η κυβέρνηση, δεν μπορεί να το κάνει μόνο η κυβέρνηση, αλλά όλοι μα πρέπει να κινηθούμε. Αυτού του είδου η προσέγγιση είναι αυτή που έχω υπόψη μου όταν μιλώ για πιο εφάνταστη προσέγγιση στην περιοχή. Και είναι ένα στοιχείο που αφορά και τη Βοσνία διότι περισσότεροι ε, πολίτες δεν έχουν τρόπο να εκφράσουν τις απόψεις τους. Οι εθνοτικές ελίτ έχουν μπλοκάρει τη διαδικασία. Αυτό ισχύει κυρίως για τη Βοσνία και είναι ένα μεγάλο εμπόδιο για τη Βοσνία αυτό. Σας ευχαριστώ. Κύριος Κωνσταντίνος Τζα... από το Ελληνικό Κοινοβούλιο έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε θα ενώσω και εγώ τη φωνή μου με όσους προλάλησαν και είπαν ότι η σημερινή σύσκεψη είναι πράγματι μια σημαντική, μια σημαντική υπόθεση που θα ασχοληθεί και θα μαζέψει, θα ενώσει όλες τις απόψεις που αφορούν ένα και μόνο ζήτημα. Το γεγονός ότι τα Δυτικά Βαλκάνια είναι ευρωπαϊκός χώρος και μέσα σε αυτό το χώρο θα πρέπει να οικοδομηθούν θεσμοί ευρωπαϊκής έμπνευσης που έχουν σαν σκοπό και προοπτική την ενσωμάτωση των λαών της βαλκανικής μέσα στο γενικότερο οικοδόμημα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Από πλευράς της Ελλάδας, όχι μόνο σήμερα, αλλά και στο παρελθόν υπήρξαν δράσεις που έχουν ενωθεί με πολύ θεμελιώδεις ιστορικές διεργασίες και αφορούν την ενοποίηση των λαών των Βαλκανίων. Πριν τα βαλκάνια μεταβληθούν σε πυρηνταποθήκη της ευρώπης είχαν προϋπάρξει χώρος συνένωσης συνεργασίας και ειρηνικής συνύπαρξης λαών που ούτε η οικονομία ούτε οι διαφορετικές γλώσσες ούτε οι διαφορετικές καταγωγές ούτε οι διαφορετικοί πολιτισμοί είχαν γίνει εμπόδιο στο να υπάρχει πολύ καλή συνεργασία μεταξύ αυτών των λαών. δυστυχώς ο 20ος αιώνας με τον τρόπο που οδήγησε την ιστορία στις ακρότητες τις γνωστές εμφάνισε το μοσαϊκό αυτό των κρατών που σήμερα έχουμε υποχρέωση να τα εντάξουμε στην κοινή ευρωπαϊκή υπόθεση. όμως δεν θα πρέπει αυτό να γίνει χωρίς αρχές και χωρίς βέβαια να λαμβάνουμε υπόψη μας τις αξίες επάνω στις οποίες πρέπει να στηρίζεται η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση τις αξίες που έχουν να κάνουν με τη δημιουργία ενός ενιαίου χώρου στον οποίο πράγματι το κράτος δικαίου οι δημοκρατικές διαδικασίες τα δικαιώματα των άλλων η πολυπολιτισμικότητα αλλά και τα συμφέροντα τα ιδιαίτερα που μπορεί να έχει ένας λαός θα πρέπει να την χάνουν του ανάλογου σεβασμού. γι' αυτό ακριβώς η ελλάδα και σε αυτή ακριβώς τη σημερινή ιστορική φάση διεκδικεί να είναι βασικός συντελεστής της ενοποίησης όλης αυτής της οικογένειας στα πλαίσια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. κυρίως όμως θα πρέπει επειδή ελέγχθη και ακούστηκε προηγουμένως να γίνει αυτή η διαδικασία με βάση βέβαια τις αρχές της καλής γειτονίας και με σεβασμό στις διαδικασίες που ήδη έχουν ξεκινήσει στα πλαίσια του οηε και αφορούν την προσπάθεια υπό την εποπτεία του γενικού γραμματέα του οηε για την εξέβρεση μεταξύ της πρώην ιουγκοσλαβικής δημοκρατίας της μακεδονίας και της ελλάδος μιας αμοιβαία αποδεκτής ονομασίας. αυτό δεν προσβάλλει κανέναν και κυρίως δεν αποτελεί μειονέκτημα για τη διαδικασία αυτής της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης των δυτικών βαλκανίων στην οποία όλοι προσβλέπουμε με πολύ μεγάλη αισιοδοξία. ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και τώρα ο κύριος ε, ναντά από τη Γαλλία, ο οποίο σας ζήτησε μπλε κάρτα. σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο Βρετανό συνάδελφο που μίλησε από το House of Lords ε, και εγώ πιστεύω, όπω και αυτό ότι η Ευρωπαϊκή ε, Ενοποίηση ήταν μια ιστορία επιτυχία και στην εμπειρία μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είδα πώς επεκτάθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση σε 27 κρατη από 12. Ήταν μια πραγματικά ιστορική διαδικασία, αξιοσημείωτη και φυσικά η διεύρυνση προς τα Δυτικά Βαλκάνια αποδέχομαι ότι θα υπάρχουν προκλήσεις, αλλά αποτελεί ένα σημαντικό βήμα και ένα δικαίωμα το οποίο έχουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες και τα Δυτικά Βαλκάνια υπό το άρθρο 49 είναι ευρωπαϊκά κρατή. Επίσης ε, πιστεύω ότι αποτελεί και την κόλλα αν θέλετε που ενώνει τις χώρες αυτές ε, στον αγώνα τους κατά της διαφθοράς της, ε, του εγκλήματος, του αγώνα τους υπέρ της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τέλος το πιο σημαντικό είναι να διατηρηθεί η ειρήνη στην περιοχή. Θυμόμαστε όλη την αιματοχυσία της δεκαετίας του 90, δεν θέλουμε να επαναληφθούν όλα αυτά και όσο και αν χρειάζεται να πείσω πολλές φορές το εκλογικό μου, την εκλογική μου περιφέρεια που είναι αρκετά σκεπτιστική ότι πρέπει να υπάρχει διεύρυνση με τα Βαλκάνια, θεωρούμε ότι θα είναι τεράστιος ο αντίκτυπος ε, σε ό,τι αφορά τις οικονομικές συνέπειες και το μεταναστευτικό κύμα προς τις χώρες μας προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα δικαίωμα. Επί του παρόντος φυσικά είμαστε κάπως επικεντρωμένοι εδώ στο Κοινοβούλιο αλλά και στα, Εθνικά Κοινοβούλια στο θέμα της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, δικαίως. Και επειδή είμαι ο σταθερός εισηγητής για το Μαυροβούνιο του Κοινοβουλίου, ακούσαμε, μάλλον συμμετέχει και εκπρόσωπος του Κοινοβουλίου σήμερα εδώ. Ίσως οι συνάδελφοί μας λοιπόν να αισθάνονται ότι τους έχουμε ξεχάσει γιατί όλες οι συζητήσεις ε, γίνονται για την Τινησία και τη Λιβύη και την Αίγυπτο και φυσικά έχουμε ευθύνη απέναντι στις χώρες αυτές. Να μην ξεχνάμε όμως και τα Δυτικά Βαλκάνια για το θέμα του Μαυροβουνίου. Σήμερα το πρωί ζήτησα από τον κύριο Λάιτσεκ να μου πει πώς θα έχουμε κάποια ημερομηνία από την Κομισιόν για την έναρξη των διαπραγματεύσεων με το Μαυροβούνιο. Είναι υποψήφια χώρα, αλλά βρίσκεται σε μια ενδιάμεση κατάσταση. Δεν έχουν συγκεκριμένη όμως ημερομηνία για την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Νομίζω ότι μετά το καλοκαίρι θα έχουν έναν πραγματικό οδικό χάρτη προς την προσχώρηση. Ξέρω και ότι ο Πρωθυπουργός ε, έχει αναλάβει προσωπικά το θέμα της ε, ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρόκειται να επισκεφτώ τη χώρα σύντομα. Επίσης, είμαι υπέρ της ε, Διακοινωνιστικής ομάδας με την Μακεδονία. Θα ήθελα να καλέσω την Ουγγρική Προεδρία να χρησιμοποιήσει ό,τι μέσα έχει στη διάθεσή της για να βρεθεί μια λύση για αυτό που για τους εξωτερικούς παρατηρητές φαίνεται ένα ε, αδιέξοδο ακατανόητο σε ό,τι αφορά την ονομασία για όλους τους άλλους από όλες τις άλλες χώρες δεν είναι λογικό όλο το μέλλον μιας χώρας σε ό,τι αφορά την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ να παρεμποδίζεται επειδή θέλουν να ονομάζονται Μακεδόνες και όχι Φάιρομ. Να καλέσω τους Έλληνες φίλους να ξανασκεφτούν για τη σταθερότητα της περιοχής ότι θα πρέπει να επιτρέψουν στην Μακεδονία ιδιαίτερα και ενώπιση των εκλογών τον Ιούνιο, γιατί οι ακραίοι, ξέρετε, αν θεωρηθούν ότι δεν τους υποστηρίζει η διεθνή κοινότητα, θα υπάρχουν ε, αποτελέσματα και συνέπειες ε, στις εκλογές. Για το θέμα του Κωσυφοπεδίου είναι λίγο ασυνήθιστο για το Ευρωκοινοβούλιο. Πάντα ήμουν υπέρ όμως ε, μιας δίκαιης κατανομής. Πώς μπορείτε να εξηγήσουμε το εξής. Αφενός το κουαρτέτο η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπέρ της ε, ειρήνης ε, για να επιληθεί. Ναι, σας ολοκληρώθηκε ο χρόνος ομιλίας σας. Ε, για την Παλαιστίνη λοιπόν και το Ισραήλ είμαστε υπέρ μιας ελληνικής λύσης, αλλά για το κοσυφοπαίδιο είμαστε κατά. Να δούμε λοιπόν αυτό το θέμα του διαχωρισμού, γιατί το πρόβλημα αυτό δεν πρόκειται να λυθεί από μόνο του. Ο κύριος Σφέραν, ο οποίος ζήτησε μπλε κάρτα. Να ακούσουμε την ερώτησή σας. Εγώ θα θέσω το ερώτημα και θα απαντήσω ποιος θέλει. Θα ήθελα να συγχαρώ την ε, Ουγγρική Προεδρία για τη σημερινή συζήτηση. Θα ήθελα εντάχει να πω στον συνάδελφο από τη Μεγάλη Βρετανία ότι η Ένωση για τη Μεσόγειο μπορεί να οικοδομηθεί κάλλιστα με περισσότερη ολοκλήρωση, δηλαδή ε, συμπερικλώντας και τα βαλκανικά ε, κράτη. Δεν πρόκειται για αντινομία. Πρώτον. Δεύτερον, μιλούν όλοι για την ενσωμάτωση των, πρώην, των δημοκρατίων της πρώην ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιτάξτε, η βασική υποχρέωση για να επιτύχει κανείς πολιτική σταθερότητα στην περιοχή εξαιρμένης της ε, προσχώρησης της Κροατίας, είναι η ενσωμάτωση της Σερβίας. Εάν δεν ενσωματώσουμε τη Σερβία ταχύτατα, δεν θα επιτύχουμε πολιτική σταθερότητα και δεν θα επικρατήσει φιλιρινικό κλίμα ε, σε όλες τις γειτονικές χώρες της Σερβίας. Είναι το πιο σημαντικό κράτος της πρώην Ιουγκοσλαβίας. Δεν μπορεί έσα ε, να επιμένουμε να πληρώνει μόνη της το τίμημα του πολέμου και δεν θα ήταν λογικό να, ε, να διεξάγουμε τις διαπραγματεύσεις υπό την αίρεση της σύλληψης αξιωματούχων που κατηγορούνται για εγκλήματα στον πόλεμο που έχει τελειώσει. Επιτέλους, θα πρέπει να αρχίσουν διαπραγματεύσεις με την Σερβία για την ένταξή της στην Ένωση. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα θα ήθελα να ζητήσω από τους ε, συναδέλφους οι οποίοι θέλουν να υποβάλουν κάποια ερώτηση, να χρησιμοποιούν κάρτα και να σέβονται το όριο του μισού λεπτού για τις ερωτήσεις ή δυνατόν. Και τώρα ο κύριος ε, Κράσνικη έχει το λόγο από το κρίσιμο παιδί. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε Μπούζεκ, αγαπητοί συνάδελφοι, επί σειρά ετών προσπαθήσαμε να στεριώσουμε τη δημοκρατία και του κράτους δικαίου στη χώρα μας. Επίση, προσπαθήσαμε να υλοποιήσουμε το στόχο της πολιτικής σταθερότητα. Βέβαια υπήρχαν ε, οι δυσκολίες από μια οικονομία που ήταν κατεστραμμένη. Όμως εμείς μπορέσαμε να κάνουμε βήματα προόδου ε, στον οικονομικό τομέα και επίση όσον αφορά και ε, το επίπεδο ζωή των συμπολιτών μα. Βεβαίω, υπήρχε το θέμα των ε, υποδομών, των υποδομών που είχαν καταστραφεί από τον πόλεμο. Εκεί επίσης καταφέραμε να προοδεύσουμε και να προχωρήσουμε σαν συγκρότηση της χώρας. Σήμερα προσπαθούμε να κατασκευάσουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο, να το ολοκληρώσουμε. Είναι ένας αυτοκινητόδρομος που θα μας συνδέει με την ε, αλβανική ακτή, αλλά και από την άλλη μεριά θα πηγαίνει προς τη Σερβία και κατά επέκταση προς την Ευρώπη. Ε, τα τελευταία χρόνια επίσης ε, έχουμε προβεί ή στην κατασκευή ενός ε, δικτύου τηλεπικοινωνιών. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι πέρα από το χέρι μας, ούτως ώστε να μπορούμε να ελκύσουμε επενδύσεις από το εξωτερικό. Επίσης, έχουμε θεσπίσει ένα σύνταγμα που παρέχει εγγύηση για τις ατομικές ελευθερίες και κατοχυρώνει και τις μειονότητες. Προσπαθούμε επομένω να χαράξουμε μια πολιτική ισότητας όλων ενώπιον των αρχών ενώπιον του νόμου. Και επίση καταβάλουμε σημαντικέ προσπάθειε ώστε να υπάρχει αγαστή συνεργασία με τι ε, γειτόνε χώρε. Επίση προσεγγίσαμε και προσπαθούμε να ενταχθούμε πλήρω ε, σε όλου του φορεί, οργανισμού, ε, θεσμικά όργανα, τα ευρωατλαντικά. Θέλουμε να προσεγγίσουμε επομένω και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, να μπορέσουμε να πετύχουμε ελεύθερη διακίνηση των ε, υπηκών της χώρας να μπορούν να κυκλοφορήσουν στην Ευρώπη χωρίς όρεση διαβατηρίων και έτσι να είναι ευκολότερη η ένταξη και η προσέγγιση. Έτσι θα μπορούμε να επισκεφτούμε ευκολότερα τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Τώρα πάντως επικρατεί κάποια απεσιοδοξία όσον αφορά την ε, άρση του καθεστώτος ε, των, των ε, θεωρήσεων στη χώρα μας. Ε, πάντως ο κόσμος αγαπά τη Δυτική Ευρώπη και επιθυμεί διακαώς ελεύθερη κυκλοφορία για πρόσωπα και εμπορεύματα και κυρίως αυτό αφορά τους νέους. Τους νέους που διψάνε για μάθηση, διψάνε για να σπουδάσουν στα πανεπιστήμια της Δυτικής Ευρώπη. Ο Πρόεδρος. Ε, το λόγο θέλει η κυρία Χερσκόφσκα από την Πολωνία. Ευχαριστώ Πρόεδρε κυρίες και κύριοι. Όσον αφορά το θέμα που συζητούμε, θα πρέπει να καταβάλουμε τις δέουσες προσπάθειες για επίλυση των προβλημάτων. Επί σειρά ετών καταβάλλονται προσπάθειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, σε διάφορες αξίες. Μία από αυτές είναι η ασφάλεια των ανθρώπων, η ελεύθερη μετακίνησή τους και η δημιουργία ενός χώρου ε, ασφάλειας, δικαιοσύνης και ελευθερίας. Οι αρχικές διατάξεις της συνθήκης αναφέρονται στις εγγύσεις που δίνει για την ύπαρξη αυτού του χώρου η Ευρωπαϊκή Ένωση για το χώρο ελευθερίας και ελεύθερης διακίνησης ατόμων και αγαθών χωρίς μεθοριακούς ελέγχους όσον αφορά τα εσωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αναφέρεται η συνθήκη και στην καταπολέμηση του εγκλήματος. Έτσι θα έχουμε μια ασφαλή αλλά ανοιχτή Ευρώπη που θα υποστηρίζει την ευμάρεια, το υψηλό βιωτικό επίπεδο των πολιτών της. Αυτός ο χώρος λοιπόν όλο και διευρύνεται και υποστηρίζει την λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Επίσης έχουμε και άλλους φορείς, την Europol και την Eurojust, που ε, ελέγχουν τις εξελίξεις σε αυτό το χώρο δικαιοσύνης, ελευθερίας Υπάρχει επίση και συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων και πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων στη διαδικασία την όλη την ευρωπαϊκή που ακολουθείται. Ο χώρο ελευθερία, δικαιοσύνη και ασφάλεια τώρα στι χώρε τη Βαλκανική είναι κάτι που αν πραγματοποιηθεί θα επιτρέψει σε αυτές τις χώρες να πληρούν ε, τις προδιαγραφές που απαιτούνται για να φτάσει στο σωστό επίπεδο. Ο διάλογος και οι επαφέ που ξεκινήσαμε θα πρέπει να επικεντρώνονται συνεχώς επί μιας ισορροπημένης δημιουργίας δυναμικού αυξήσεως των δυνατοτήτων του δικαστικού τομέα. Θεωρούμε ότι η σταδιακή ένταξη των υποψηφίων χωρών και των άλλων χωρών που θέλουν να θέσουν υποψηφιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα αυξήσουν τη σταθερότητα στην περιοχή. Η πρόοδο για την ένταξη σε αυτέ τι χώρε εξαρτάται όμω και από την ενίσχυση που μπορούμε να του δώσουμε. Τι μέσα μπορούμε να του διαθέσουμε για να υποστηρίξουμε του πληθυσμού στα θέματα πολιτισμικά και παιδεία. Η... Θα αναλάβει το επόμενο εξάμενο η Πολωνία την Προεδρία τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω και κοιτάμε και μαθαίνουμε από την Ουγγρική Προεδρία και προσευχόμαστε ε, οι ενταξιακέ διαπραγματεύσει να συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της Πολωνικής Προεδρίας να ενταχθεί η, Πολωνία, ε, ενταχθεί η Κροατία συγγνώμη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο, κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θέλω να πω ότι θεωρώ σημαντικότατο το ότι η Ουγγρική Προεδρία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλιο που επέλεξαν ακριβώς αυτό το θέμα. Δηλαδή τα Δυτικά Βαλκάνια και νομίζω ότι σαν μέλος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα ήθελα να υπογραμμίσω το ότι η δική μας δουλειά ακριβώς γίνεται ούτως ώστε οι νέοι να ε, καταλάβουν ότι μπορούμε να βλέπουμε τα καθημερινά προβλήματα τους, τα προβλήματα των νέων στην Ευρώπη και γι' αυτό η απελευθέρωση από το καθεστώς ε, θεωρήσεως διαβατηρίων είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι έτσι θα μπορούν οι νέοι να έχουν πρόσβαση στην Ευρώπη ταξιδεύοντας από αυτές τις χώρες και ε, έχουμε υπόψη μας και τις μελλοντικές γενιές ε, έτσι θα αλλάξει η νοοτροπία τους και θα αλλάξει η νοοτροπία τους και στη χώρα τους όταν επιστρέφουν. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα και βλέπουμε κάποια προβλήματα σε αυτή τη φάση τα οποία έχουμε την εντύπωση ότι ε, θα ήταν ανεπίλητα, αλλά με αυτό που προανέφερα θα μπορούσαμε να λύσουμε τα προβλήματα. Δεν υπάρχει ανάγκη θεώρηση. Αν μπορούν να ταξιδεύουν ελεύθερα, αν μπορούν οι νέοι να, ε, να, να βλέπουν τι γίνεται στην Ευρώπη, πώς σκέφτεται ο κόσμο στην Ευρώπη. Έτσι μπορεί να τους επηρεάσει η Ευρώπη στην καθημερινή του ζωή. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο εκπρόσωπο τη Κροατία. Η κυρία Ντομπράφσκοβιτς έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, να ευχαριστήσω την Ουγγρική Προεδρία που διοργάνωσε το συνέδριο αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψη. Και σε αυτή την ευκαιρία θα ήθελα να πω ότι ανυπομονώ, όχι μόνο εγώ προσωπικά, αλλά όλοι μας ε, στην Κροατία, να βάλουμε ένα τέλος στις διαπραγματεύσεις μας ε, μέχρι το τέλος ε, της Ουγγρικής Προεδρίας, μέχρι το τέλη Ιουνίου. Θα πρέπει να πω εδώ ότι είμαστε πρωταθλητές στην περιοχή για τη διαπραγμάτευση επί έξι χρόνια. Ελπίζω να τερματιστεί τέλη Ιουνίου η διαδικασία αυτή με την υποστήριξή σας. Θα ήθελα να υποστηρίξω τον ε, πρόεδρο του Κοινοβουλίου μας, ο οποίος τόνισε ότι ε, δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην περιφερειακή συνεργασία. Όπως θα γνωρίζετε, η Κροατία αναγνωρίζεται ως ηγέτης της περιοχής. Μία, ένα αποδεκτικό στοιχείο είναι ότι ο υπουργό μας υπέβαλε μετάφραση της νομοθεσίας της για να βοηθήσει το Μαυροβούνιο και τη Σερβία προς την ευρωπαϊκή τους κατεύθυνση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας να καταδείξουμε ότι υποστηρίζουμε και προωθούμε την περιφερειακή συνεργασία και το νομοθετικό πλαίσιο επίσης αποτελεί προτεραιότητά μας. Να ξέρετε ότι έχουμε περάσει πιο πολλούς από 520 νόμους στο κοινοβούλιο μας γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι χωρίς ανθρώπινα δικαιώματα, χωρίς κράτος δικαίου, χωρίς δημοκρατικό πλουραλισμό, χωρίς όλα αυτά τα στοιχεία δεν υπάρχει ελεύθερη αγορά, δεν υπάρχει οικονομική ανάπτυξη. Το θέμα της ε, συνεδρίασής μας είναι η οικονομική ενσωμάτωση. Προσπαθούμε να συμβάλλουμε στην οικοδόμηση υποδομών στην περιοχή μας. Προσπαθούμε να συνδράμουμε στην οικοδόμηση ε, διαδρόμων όπως ο 5C για την σύνδεση με την Νότια Αδριατική και επίσης κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε την ε, οδό Αδριατική, Αδριατικής Ιωνίου. Γιατί χωρίς αυτήν δεν θα είναι δυνατή η οικονομική ανάπτυξη, τηρώντας ε, αυστηρά τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Να σας ε, διαβεβαιώσω ωστόσο ότι έχουμε σχεδόν συμμορφωθεί με όλα. Δεν θέλουμε λοιπόν να καταστεί αυτό πολιτικό ζήτημα. Σας ευχαριστούμε που μας ε, ενθαρρύνετε σε ό,τι αφορά την ε, ένταξή μας στην Ένωση, σε ό,τι αφορά την στρατηγική επικοινωνίας. Κάποιος το έθεσε το ερώτημα αυτό. Υπάρχει τέτοια στρατηγική επικοινωνίας ε, στην Κροατία και είμαι βέβαιη ότι οι πολίτες μας θα ψηφίσουν ναι. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Και τώρα έχουμε ένα τελευταίο μιλητή, τον κύριο Βλαντιμίρ Τόσεφ από τη Βουλγαρία. Господин Κύριε Πρόεδρε, έχουμε τις προοπτικές, τις ευρωπαϊκές για τα Δυτικά Βαλκάνια που θα αποτελέσουν εγγύηση για την επίτευξη ειρήνης και σταθερότητα στην περιοχή. Παρακαλούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσέξει περισσότερο την περιοχή μας, περισσότερο τα Δυτικά Βαλκάνια, διότι πρόκειται για μια περιοχή που σημαίνει πολλά για την ασφάλεια όλη τη Ευρώπη. Πάρα πολύ θετικό το ότι όπου να ολοκληρωθούν θετικά θα ευοδοθούν οι α, επαφές με την ε, Κροατία. Πάρα πολύ σωστό θα είναι το μήνυμα το οποίο θα ε, σταλεί σε όλες τις χώρες εάν επομένως ε, ολοκληρωθεί η προσχώρηση της Κροατίας. θα πρέπει να συνεχίσει την πορεία της Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και θα πρέπει και η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας να εφαρμόσει ε, τις αποφάσεις ε, της 14 Δεκεμβρίου του 2010 ε, γιατί το Συμβούλιο τότε είχε αποφανθεί όσον αφορά τα της προσχώρησης και της φοράς εκείνης. Βεβαίως θα είναι πάρα πολύ κρίσιμα τα αποτελέσματα των εκλογών που θα γίνουν σύντομα η χώρα θα μπορέσει επομένω με την νέα κυβέρνηση να επικεντρώσει περισσότερε προαθειέ στην ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να ε, γίνει η κύρωση των ε, συμφωνιών που αφορούν την ε, σύνδεση, την προσέγγιση Ερδίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πρέπει να διεξέλθει και την αίτηση της χώρας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά για την Σερβία αλλά και για την ευρύτερη περιοχή. Εμείς θεωρούμε ότι η αξιολόγηση του Επιτρόπου Φιούλε ε, που έγινε το 28 Μαρτίου ε, ήταν ο καταλήτης ε, που επετάχυνε τις διαδικασίες προσέγγισης της χώρας. Όσον αφορά το κατά πόσο θα πληρούνται τα κριτήρια της Κοπενχάγης, αυτό θα αποτελέσει επίσης ένα πλεονέκτημα για την ένταξη της χώρας. άνοιξαν πάρα πολλοί φάκελοι ούτως υπήρουν που εκκρεμούσαν στη χώρα και ούτω ώστε να φύγουν όλε οι σκιές που βάρναν την πολιτική ιστορία. Επομένω, με την προσχώρηση θα γίνουμε και εμεί μέλο τη ευρωπαϊκή οικογένεια και αυτό θα είναι πάρα πολύ θετικό για την χώρα. Έτσι θα αποδειχθεί ότι μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Και ακόμα πιο δύσκολο. Τόσο αφορά την Αλβανία. Η Αλβανία θα πρέπει να καταφέρει ε, να πληρεί τα κριτήρια της Κοπενχάγης. Θα πρέπει να δούμε το πώς τη χειραγώγηση της ιστορίας θα την αφήσουμε πίσω μας, στο χρονοτούλαπο. Και έτσι να προχωρήσουν, μπορούν τα Δυτικά Βαλκάνια να προχωρήσουν για να μπουν σε Ευρώπη. Σας, σας ευχαριστούμε. Δεν έχουμε πλέον χρόνο στη διάθεσή μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν στη συζήτηση και παραδίδω τις κοιτάλες στον Συμπρόεδρο, τον κύριο Θα ήθελα να σας ενημερώσω για κάτι. Τις ε, προσεχείς δύο ώρες θα συνεχιστεί η συνεδρία σε δύο διαφορετικές ομάδες εργασίας. Η πρώτη ομάδα εργασίας εργασίας-συνεργασία στον τομέα της ελευθερίας, τη δικαιοσύνης και της ασφάλειας. Θα συνεδριάσει εδώ η πρώτη ομάδα εργασίας. Δεν χρειάζεται να μετακινηθείτε. The ε, θα καλύψουμε τα σύνορα, τις θεωρήσεις, τα μεταναστευτικά ζητήματα καθώς και την αστυνομική και δικαστική συνεργασία. Η κυρία Κόπα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η κυρία Εύα από το πολιτικό Κοινοβούλιο θα συμπροεδρεύσουν. Η κυρία Ντορισπάκη είναι συγγήτρια. Δεύτερη ομάδα εργασίας, ε, ενσωμάτωση ένταξη των πολιτών. Στην 3 σε 50 θα συνεδριάσει ε, η δεύτερη ομάδα εργασία. Είναι στον ίδιο όροφο, στο ίδιο κτίριο προφανώ, ακριβώ απέναντι. Μόλι βγείτε από την αίθουσα, απέναντι ακριβώ. Είναι πάρα πολύ εύκολο να το βρείτε. Ο στόχο είναι να εξετάσουμε την πολιτιστική ποικιλομορφία, τη συμβουλή πολίτης της παιδείας στη διαδικασία ένταξης των χωρών Δυτικών Βαλκανίων στην Ένωση, η κυρία Ζακλίν Γκαλάν. Από την Βελική Βουλή των Αντιπροσώπων και ο κύριος Κάτσιν, ευρωβουλευτής, θα συμπροεδρέψουν Ο κύριος Μιχάλη Μπάλα είναι ο εισηγητής από την Ουγγρική Εθνοσυνέλευση. Οι ομάδες εργασία πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τι συζητήσει τους μέχρι τις 7 το βράδυ. Μετά μεσημβρίας, όχι προ, μετά, σε δύο ώρες από τώρα. Τα πιο σημαντικά πρόσωπα, οι πιο σημαίνουσες φυσιογνωμίε είναι οι εισηγητέ. Ζητώ συγγνώμη που σας το λέω. Γιατί το λέω όμω αυτό θα σα εξηγήσω. Καλείστε να παρουσιάσετε αύριο το πρωί στην Ολομέλεια τις εκθέσεις που θα προετοιμάσετε και θα μοιραστούν σε όλου του συμμετέχοντες οι εκθέσεις σας. Θα θέλαμε λοιπόν να συντάξετε μία έκθεση μετά το πέρας των συζητήσεων ή στα αγγλικά ή στα ε, γαλλικά κατά προτίμηση αλλά προφανώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποια γλώσσα θέλετε και θα μεταφραστεί αμελητή το κείμενο. Στις 7, κοκτέιλ. Κατόπιν ε, δείπνο με μπουφέ. Στο Γεχούντι Μενοχήν είναι ένας χώρος στο ίδιο κτίριο, αλλά στον πρώτο όροφο. Πρέπει να κατεβείτε δύο ορόφους. Και θα το βρείτε. Πάρτε και το ασανσέρα, αν θέλετε. The invitation card for the dinner and information about the location of the... Επίσης, ε, στους φακέλους που σας μοιράσαμε έχετε όλες αυτές τις πληροφορίες. Δεν χρειάζεται να τις απομνημονεύσετε. Σας ευχαριστούμε για τη σημερινή συζήτηση εσάβριον στην Ολομέλεια και θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως στις 7 για το κοκτέιλι και μετά για το δείπνο. Ευχαριστώ.